Meine Κυρίες και κύριοι, σας ε, καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία ε, ημιμερίδα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις και στη, με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Προτού όμως ασχοληθώ με την επίσημη ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να εκφράσω και φαντάζομαι ότι είναι εν ονόματι σας ότι όλοι έχουμε ταραχθεί και συντριβεί από την κατάσταση η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία. Έχουμε συνεχείς ανακοινώσεις και εκεί που νομίζουμε ότι πέρασε το χειρότερο έχουμε και καινούργιες ε, εξελίξεις που δείχνουν ότι δεν διαβλέπεται το τέλος αυτής της κατάστασης. Θα παρακαλούσα λοιπόν εν ονόματι της ε, ε, συμμετοχής μας να σηκωθούμε για ενός λεπτού σιγή. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Ich Καταρχήν ε, θέλω να χαιρετήσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι τόσο συχνό να έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες, και χαίρομαι που ε, ήρθατε τόσο πολύ άριθμοι ανταποκρινόμενοι στις, ε, στην πρόσκλησή μας. Έχουμε 18 ε, κοινοβούλια που εκπροσωπούνται και πολλές φορές και από τα δύο σώματα της Εθνικής Βουλής. Παρακαλώ λοιπόν να σχολιάσετε τα θέματα που έχουμε προς συζήτηση αλλά ε, το ερωτηματολόγιο ως επτοπλίστων έχει ε, απαντηθεί. Ξέρετε ότι ε, η Επιτροπή Κρίς καταρτίστηκε στο τέλος του 2009 και ασχολήθηκε καταρχήν με τους λόγους, τις αιτίες της κρίσεως και προσπάθησε να διατυπώσει συστάσεις για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, θέλω όμως να κάνω μία σύντομη ε, σύνοψη διότι διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και αν δεν ακολουθήσουμε στα επόμενα έτη τη σωστή οδό τότε κινδυνεύουμε ε, να μην μπορέσουμε να επανέλθουμε στο status quo άντε πριν την κρίση αλλά να βρεθούμε σε δυσμενέστερη κατάσταση και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα υπόλοιπα σώματα όπως το G20 ο ΙΕ πρέπει να εκπροσωπείται από ένα άτομο και να μιλάμε μία φωνή. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ισχυρή επιτροπή και μία, έναν ισχυρό επίτροπο που να είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Και αυτό διαπιστώβουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές συναντήσεις για να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις παρόλο που εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια καλούνται εκ των υστέρων απλώς να προσυπογράψουν τις αποφάσεις. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει όλο και πιο έντονος ανταγωνισμός και πρέπει να προωθηθεί η υποδομή και αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία για να κάνουμε όλοι μαζί αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιο κράτος μόνος του όπως στην ε, ψηφιακή Ευρώπη, ε, την διοικητική μέρημνα, τις ε, συγκοινωνίες και μεταφορές και ούτω καθεξής. Και αυτές οι διαρθρωτικές δομές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά ομόλογα και αυτό θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Και τέλος πρέπει να καταφέρουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ε, μέση ε, τάξη ε, και να την αναπτύξουμε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να παραμείνει στη θέση του και εδώ δεν επαρκούν τα ευχολόγια, χρειαζόμαστε πράξεις. σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο του διαλόγου στο, τον οποίο διεξάγουμε εδώ και μερικούς μήνες με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό και όπως σας είπα χαίρομαι ιδιαιτέρως ότι παρίστανται εδώ τόσο οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων καθότι προσπαθήσαμε να ε, ε, διατυπώσουμε μία ίδια γνώμη με εκπροσώπους των Κοινοβουλίων και των, ε, και των χωρών πήγαμε στην Τσεχία, στην ε, Ισπανία, στη Γερμανία και την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε στην Αθήνα κατά τρόπον ώστε να ε, ε, διαπιστώσουμε ποιες είναι οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε δύο θέματα. Στο πρώτο ήμιση θα εξετάσουμε τις αναγκαίες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση διότι αν δεν εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε τις κρίσεις και να μειώσουμε τα, τα χρέη μας το οποίο ε, επιβάλλεται. Η δεύτερη συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις ε, ενέργειες που πρέπει να αναλυθούν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής ε, του 2020 διότι η στρατηγική της Λισαβόνας είχε προβλέψει ότι η Ευρώπη έπρεπε ε, να προχωρά γρήγορα και να γίνει ηγετική διεθνώς αλλά απέτυχε. Ο πρώτος μιλητής μας σήμερα κάθεται αριστερά μου είναι ο Τόμας Μύρο, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης από το 2008 και αυτός τα, τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει τη δυναμικά την τράπεζα, την έχει κατευθύνει διαμέσου της κρίσεως και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο όγκος τον οποίο έχει επιτύχει σε πιστώσεις η τράπεζα και σε χορηγήσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τις ενάρξεώς της με 9 δισεκατομμύρια. Προηγουμένως ε, ήταν ε, ε, υφυπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο και νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ χρήσιμος για μας όχι μόνο σαν δημόσιος λειτουργός αλλά διότι έχει υπάρξει και σε δύο φάσεις πολιτικός περιμένουμε να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία του και στη συνέχεια θα έχουμε σχόλια επί του θέματος καταρχήν από την Τρόικα, την ε, Τριημερή Επιτροπή της προηγουμένης, ε, της Βελγικής δηλαδή, της προηγουμένης ε, της ε, ε, Ουγγρικής, της επομένης της Πολωνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έτσι επί 18 μήνες υπάρχει μία συνέχεια, άρα πρώτα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων αυτών των τριών χωρών και μετά οι εθνικοί ε, εκπρόσωποι και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μύρο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με καλέσατε και για την εισαγωγή που κάνατε. Είναι προνόμιο για μένα να ανταλλάζω απόψεις μαζί σας που είσαστε εκπρόσωποι των ε, πολιτών της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Με τα χαρά μοιράζομαι την πρόσκληση με τον πρόεδρο Μάιστα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τον οποίο υπέγραψα μόλις τώρα μια νέα συμφωνία γενική συνεργασίας που συμπεριλαμβάνει σαν τρίτο εταίρο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω το ότι έχετε αφιερώσει πολύτιμο χρόνο για να ασχοληθούμε με ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που αντιμετωπίζουμε αυτή την εποχή και αυτό είναι αποδειγμένο, δηλαδή πώς να ξαναζωγονήσουμε την πραγματική οικονομία και πώς θα χρησιμοποιηθεί σαν κινητήρας μιας βιώσιμης ε, ανάπτυξης με γρήγορους ρυθμούς. Όπως γνωρίζετε, η οικονομία της Ευρώπης πέρσι επανήλθε στην ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της βελτίωσε την εκροή της κατά 1,8% το προϊόν της το 2010 όμως ε, σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας απομένει και προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ευρωζώνη συνεχίζονται. Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές ε, προκλήσεις και η ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από εξωτερικές εξελίξεις στις ε, προχωρημένες οικονομίες και από την τιμή των διαφόρων βασικών αγαθών. Όμως υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο παραμένει αυτή η ανησυχία. Υπάρχει το δυσάρεστο συνέστημα, η ανησυχία, ότι πολλές ε, αδυναμίες που εξετέθησαν από την κρίση δεν ε, έχουν ε, διορθωθεί. Και είναι κατανοητό ότι αυτό ήταν ανέφικτο όταν ήταν στην ακμή της η κρίση. Όμως τα επόμενα χρόνια θα είναι κρισίμου σημασία ώστε να κινηθούμε προς ένα μοντέλο πιο στέρεο, αναπτυξιακό μοντέλο. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, τρεις τομείς έχουν ύψη τη σημασία. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναζωογονήσει την μακρά και περήφανη παράδοση της κατασκευής προϊόντων υψηλής ποιότητας. Όμως οι οικονομίες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στο χρηματοστατικό τομέα, στις οικοδομές και τις υπηρεσίες. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει την τεχνολογία εχμής της και θα πρέπει να επενδύσει μεγάλα ποσά σε ένα εργατικό δυναμικό που θα είναι καλά εκπαιδευμένο, έχοντας σαν στόχο μια πολύ ανταγωνιστική προσέγγιση που θα μπορέσει αυτή η προσέγγιση να χρησιμοποιηθεί σαν κινητήρας ε, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Απαιτείται να γίνουν εσωτερικές αλλαγές σε κάθε χώρα και πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Αρκετά κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ένα πρόγραμμα που ακόμα συμπεριλαμβάνει ατέλειωτες μεταρρυθμίσεις όπως είναι η ιδιωτικοποίηση και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αυτά μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και μπορούν να αναζωογονήσουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Πολλά από αυτά τα θέματα ίσως να μπορούν να εφαρμοστούν οι προσεγγίσεις και σε δυτικά κράτη-μέλη. Πέραν αυτού, η ενή αγορά πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, ούτω ώστε το συγκριτικό όφελος διαφόρων χωρών να χρησιμοποιηθεί ε, με την πρόοδο της οικονομικής ολοκλήρωσης. Οι εναπομένοντες φραγμοί ε, υπάρχουν ακόμα, δεν είναι πολύ μεγάλοι, αλλά παίζουν το ρόλο τους. Μερικά παραδείγματα. Η Οδηγία Περιπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ακόμα εξαιρεί ένα ευρύ φάσμα τομέων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιλογής στα πλαίσια εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου και πόρο απέχουμε από μια πραγματική ενιαία αγορά. Η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων και των πανεπιστημιακών πτυχίων, των πτυχίων της παιδείας είναι σε περιορισμένο βαθμό που εφαρμόζεται και περιορίζεται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Και τρίτον, στην Ανατολική Ευρώπη επιχειρήσεις πολύ συχνά έχουν πρόβλημα για να προσαρμοστούν στο διαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε κάποιους τομείς ε, έχουν πρόβλημα και οι ίδιες οι δημόσιες αρχές να συμμορφωθούν με τις επιταγές Ευρωπαϊκής Ενώσης με τα σωστά κίνητρα, Φερρυπίν, με ένα καινοτόμο φορολογικό σύστημα που ε, τιμωρεί τη βλάβη στο περιβάλλον και τη σωστή προσέγγιση για την απασχόληση, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα για να προωθήσουμε καινοτόμα ε, παραγωγή τεχνολογίας εχμής. Θα πρέπει μετά να επανακαθορίσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα Μία συνέπεια της κρίσεως ποια είναι. Θα εισαχθούν νέες ρυθμίσεις και μηχανισμοί εποπτικοί για την ενίσχυση του τομέα. Η Βασιλεία 3 θα αυξήσει τις κεφαλουχικές απαιτήσεις και έχει σαν στόχο να ληφθούν μέτρα κατά ε, της ανάληψης πολύ μεγάλων κινδύνων. Αυτά είναι ευπρόσδεκτα βήματα. Στην Ανατολική Ευρώπη η ενίσχυση των χρηματοστικών συστημάτων σημαίνει επίσης να μάθει κανείς τα σωστά μαθήματα από τον πόνο που δημιούργησαν ε, οι, οι, οι λήψεις δανείων, οι δανειοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα από τα δύο. Ή να εφαρμόσουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και μεταρρυθμίσεις ούτω ώστε να μπουν οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη είτε εκείνοι που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μπουν στην Ευρωζώνη να αναπτύξουν αγορές σε τοπικό νόμισμα και να μετακινηθούν προς δανειοδότηση στο τοπικό συνάλλαγμα, στο τοπικό νόμισμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι ο χρηματοστικός τομέας θα ξαναγίνει υπηρέτης της πραγματικής οικονομίας και όχι ένα σύστημα ε, που έχει σαν αφορά τον εαυτό του και είναι αυτός σκοπός. Λοιπόν, είναι ένα ένιγμα που δεν έχει επιληθεί ακόμα. Η παγκόσμια αγορά για τα παράγωγα έχει αναπτυχθεί πέραν κάθε λογικής αναλογίας. Υπάρχουν ανισορροπίες όλων των ειδών και αυξάνονται εκ νέου αυτές οι ανισορροπίες. Οι ισχυρές δεσυνοριακές ρυθμίσεις και υποπτία απαιτούνται για να ενισχυθεί η αντίσταση του συστήματος και να εξασφαλιστεί ότι πραγματικό τομέα και επιχείρηση του πραγματικού τομέα θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και τρίτον, να πρασινίσει η οικονομία. Όσο αναπτύσσεται και βγαίνει την κρίση η ευρωπαϊκή οικονομία με νέα καινοτόμα προϊόντα και έχει την ευκαιρία μπροστά τη να απομακρυνθεί από διάφορε μορφέ παραγωγή που είναι επιβλαβεί για το περιβάλλον και μορφέ κατανάλωση που είναι επιβλαβεί. Η οικονομική κρίση μας οδηγεί στο να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κλίμα. Σε πολλές περιο... χώρες της περιοχής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Αναπτύξεως βλέπουμε ότι χρειάζονται νέες τεχνολογίες που κοστίζουν. Αλλά πολύ συχνά τα ωφέλη όσον αφορά την αύξηση παραγωγικότητας και διάφορες οικονομίες που γίνονται ξεπερνάνε τις επενδύσεις που χρειάζονται. Θα έχει μεγαλύτερο κόστος Ανατολική Ευρώπη αν δεν προσαρμοστεί στην κρίση και δεν θα μειώσει τους κινδύνους που δημιουργούνται για το κλίμα, αλλά θα βλάψει και την ανταγωνιστικότητά της η Ανατολική Ευρώπη και σε μεγάλο βαθμό, αν τα λάβει τα νέα μέτρα. Μια τέτοια αναπτυξιακή στρατηγική χρειάζεται και μεγάλες ε, επενδύσεις και το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι πώς να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα μέτρα. Και μάλιστα τώρα που εφαρμόζονται οδυνηρά μέτρα λιτότητας που κρατούν και μεγάλο χρονικό διάστημα ίσως μπορεί η εμπειρία της τράπεζας να δείξει κάποιο δρόμο που να ακολουθήσουμε. Αυτό που κάνουμε εμείς στην τράπεζα είναι να κινητοποιούμε χρήματα ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην περιοχή που καλύπτουμε και για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η τράπεζά μας έχει υποστηρίξει τη Volkswagen με την πρώτη προσπάθεια που έκανε να κατασκευάσει αυτοκίνητα στη Ρωσία αλλά ταυτόχρονα δώσαμε τη δυνατότητα σε πολωνική εταιρεία όπως είναι η Balinec να παράγει ε, σανίδες ε, και κασόνια κλπ. για να εξάγει στην Ουκρανία. Γιατί γινόμαστε ελκυστικοί όσον αφορά του επενδυτέ, έχουμε πόρους και μπορούμε να τους διαθέσουμε όχι ανταγωνιζόμενοι τους ιδιωτικούς δανειοδότες, αλλά όταν δεν υπάρχουν ε, πόροι άλλοι και μπορούμε να μοιραστούμε με τους εμπορικούς εταίρους τους κινδύνους και να ε, εντάξουμε αυτούς τους κινδύνους στον ισολογισμό μας. Και έχουμε ιστορικών συνετής διαχείρισης, σωστής αντιμετώπισης των κινδύνων και συντηρητικής οικονομικής προσεγγίσης όσον αφορά τα λογιστικά μας. Αυτά είναι θεμέλια. Μας εξυπηρέτησαν πάρα πολύ καλά. Επενδύσαμε σε πολύ φιλόδοξα έργα που βοήθησαν να αλλάξουν την οικονομία αλλά μόνο μετά από διεξοδική ανάλυση των κινδύνων. Το κάναμε αυτό. Αναλαμβάνουμε εμπευθυνότητα κινδύνου που δημιουργούν θέσει απασχόληση και μια βιώσιμη ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία. Αυτό μα επέτρεψε να ανταποκριθούμε στην ε, χρηματοστική κρίση με αποφασιστικό και γρήγορο τρόπο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει, φερειπίν στην Αίγυπτο και ενδεχομένω αλλού σε άλλε περιοχέ τη Βόρεια Αφρική, αν οι μέτοχοί μα θέλουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι το μοντέλο βαθμολόγηση ενός θεσμικού οργάνου που βαθμολογεί που βαθμολογείται με 3α και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανοικοδόμηση μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο του χρηματοστικού τομέα εν γέννη, αν αυτό ο φορέα θα πηγαίνει πολύ καλά. Όμω η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη βασίζεται σε ένα γενικότερο μάθημα που πιστεύω ότι σχετίζεται, μάλλον είναι χρήσιμο και για τις κυβερνήσεις και για τους άλλους οργανισμούς που εφαρμόζουν στόχους του δημόσιου τομέα. Ποιο είναι το μάθημα αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Ότι όλο και περισσότερο σπανίζουν οι δημόσιοι πόροι, οι κατοικοί πόροι. Και αυτοί οι πόροι που σπανίζουν θα πρέπει να συμπληρώνονται επιτυχώς από ιδιωτικούς πόρους, ούτως ώστε να επιτευχθεί αν επιτευθούν οι στόχοι της κρατικής πολιτικής, της δημόσιας πολιτικής, πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα. Ούτως ο ιδιωτικό τομέας να κινητοποιηθεί σε δραστηριότητες που είναι επωφελείς για την οικονομία στο σύνολό της. Αυτή η προσέγγιση επιφέρει δύο ωφέλη. Πρώτον, ίσως να βοηθήσει το δημόσιο τομέα θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους κρατικούς σκοπούς βγάζοντας και κέρδος. Πέρσι 1,4 δις είχαμε κέρδη. Πιο σημαντικό ακόμα, η προσέγγιση τράπεζά μας στην οικονομική ανάπτυξη εδράζεται επί της εξής υποθέσεως, ότι είναι καλύτερο κανείς να χρησιμοποιεί την ευφυΐα του ιδιωτικού τομέα για να βρεθούν λύσεις ευφυΐς που εξοικονομούν δαπάνες για να επιτευθούν δημόσιοι στόχοι από ότι ο δημόσιος τομέας να κινείται μόνος του ή ακόμα χειρότερα να κινείται σε ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να απαιτεί κάποια δημόσια χρήματα ακόμα, αλλά τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ συνετά, ούτω ώστε να μπορούμε να αποδίδουμε, να διατηρούμε το κεφάλαιο όμως πάνω από 5 δις. Το συνολικό μας κεφάλαιο που έχουμε μέχρι τώρα είναι 13 δις ευρώ περίπου. Λοιπόν, τα μέσα που έχουμε για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι συγκεκριμένα. Και χαρακτηρίζουν μια αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτό ισχύει και για τη συγχρηματοδότηση μετέρους του ιδιωτικού τομέα και αφορά και επενδύσεις σε έργα και προγράμματα του ιδιωτικού τομέα. Όμως, πιστεύω ότι αυτή η γενική αρχή ξεπερνά τα όσα κάνουμε εμείς και μόνο. Οι κυβερνήσεις έχουν μοχλούς πολιτικής για να εφαρμόσουν το πόσο επικερδής είναι η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα και αυτό το επιτυγχάνουν μέσω ρυθμιστικών εργαλείων και φορολογικών μέσων. Στον τομέα των πράσινων επενδύσεων πρωταρχικό παράδειγμα είναι σωστά ισορροπημένη τιμή για τον άνθρακα. Ο ιδιωτικός τομέας και εσείς που διαμορφώνετε την πολιτική και είστε νομοθέτες έχετε σημαντικό ρόλο να παίξετε εδώ. Οι αποφάσεις σας μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό μπορεί να ενθαρρύνει ανάληψη κινδύνων με υπεύθυνο τρόπο για βιώσιμη ανάπτυξη αντί να δίνονται κίνητρα που οδηγούν σαν ανεύθυνη ανάληψη κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες καταστροφές χρηματοπιστωτικές, ίσως και ακόμα χειρότερες από αυτές που ζήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Μύρο για αυτή την εισαγωγή και τώρα ερχόμαστε στις συνδρομές και τα σχόλια των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου ε, και το προχωρώ γαλλικά. Διαπιστώνω ότι ο κύριος Ζακ ε, Ντελόρ ήρθε πριν από λίγα λεπτά. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας καλωσορίζω. Ο κύριος Ζακ ε, Ντελόρ είναι ο μιλητής μας απόψε και γνωρίζουμε ότι είναι το άτομο το οποίο όντως προώθησε την εσωτερική αγορά και γι' αυτό χαιρόμαστε που είναι μαζί μας σήμερα και που θα μας μιλήσει το βράδυ. Τώρα όμως ξεκινάμε τη συζήτηση του πρώτου μέρους που μας έκανε μία τόσο καλή εισαγωγή ο κύριος Μύρο και καταρχήν ε, παρακαλώ τον εκπρόσωπο της, ε, ε, της Ουγγρικής Προεδρίας Έκερς μετά της Βελγικής Προεδρίας Λούξ και μετά τον κύριο Κλάινα ο οποίος είναι εκπρόσωπος της επομένης Πολωνικής Προεδρίας. Τρία λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ ακολουθήστε το παράδειγμα του κυρίου Μύρο και μην υπερβαίνετε το χρόνο σας για να μπορέσουμε μετά να έχουμε και τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών που θα έχουν μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. και καλωσορίζω όλους σας ε, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το θέμα αυτό για μας, για την Υπουργική Προεδρία, για την Ουγγαρία. Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαραίτητο μέσα από την ανάπτυξη να αμβληθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί και η απασχόληση. Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση αναδιάθρωσης σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με την στρατηγική το 2020 που θα εξελιχθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά θα είναι όλο και πιο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να μην αφήσει να χειροτερεύσει αυτή η κρίση. Όπως είπε και ο κύριος Μύροφ, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση αυτή να μιλήσει με μία φωνή. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βρούμε όλα αυτά τα σημεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στην σταθερότητα την οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη ανεργία, να υποστηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρήσης, να διευκρινίσουμε τα θέματα ε, περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά επίσης σημαντικό είναι και το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζόμενων, αλλά και η απασχόληση όσο βρίσκονται σε θέσεις περιθωριακές στην κοινωνία και σε θέματα προϋπολογισμού τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να αγγιηθούμε μια πιο αποτελεσματική μεταφορά. Κατά τη διάρκεια της Εγκουρικής Προεδρίας ε, θέλουμε να τοποθετηθούμε σε όλους αυτούς τους τομείς προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητες αυτές πραγματικά θα προωθηθούμε παράλληλα. Υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες εκείνες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της, ε, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης του 2020, και αποτελεσματικότητα, προστασία του περιβάλλοντος, θέματα διαχείρισης υδάτων, αυτό το θέμα καθίσταται όλο και πιο σημαντικό, καθότι υπάρχει λειψητρία σε όλο και πιο πολλά μέρη στον κόσμο και φυσικά θα πρέπει να διευκρινιστεί ε, τι θα γίνει με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με έρευνα, ανάπτυξη. Όλα αυτά τα θέματα και η καινοτομία ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η χρηματοδότηση όλων αυτών των τομέων. Επίσης, ε, σημαντικό θέμα θα είναι η κατανομή της ε, περιφερειακής ενίσχυσης. Αυτό περιλαμβάνει και την ΚΑΠ και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαπρόθεσμη σταθερότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Λίξ. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Μάκρο, μάικρο. Voilà. Mr. Chairman, Mr. Πρόεδρε, κύριε Μύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Πρωτού συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξη του Βελγίου για τις σημαντικές συμβάσεις, ε, συμφωνίες που συνήφθησαν το Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπαρόσο, τον κύριο Φαρόμπαϊ, αλλά και τους εθνικούς ηγέτες που με πολύ ε, κατάλληλο τρόπο κατέληξαν σε συμφωνίες για τη διασφάλιση της οικονομίας μας και του κοινωνικού μας μοντέλου. Όπως πάντα υπήρξε ευρεία συνένεση από όλες τις πλευρές ε, στα εθνικά κοινοβούλια ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μελλοντικού κοινωνικού ε, προτύπου. Να συνεχίσω στο Ολλανδικό τώρα και να μιλήσω για τέσσερα ζητήματα. Καταρχάς, πρόεδρε, ε, συνάδελφοι, έχουμε πολιτικό καθήκον να φροντίσουμε ότι μια τέτοια τραπεζική κρίση δεν θα ξαναεπανελειφθεί οι σημερινοί και οι μελλοντικοί φορολογούμενοι πληρώνουμε το παραπάνω το τίμημα της ευρωπαϊκής κρίσης. Και αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από αυτούς που χαράσουν την πολιτική είναι να ελαχιστοποιήσουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τους κινδύνους. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να επαναλάβω κάποιες αρχές που επαναλήφθησαν και σε μία βελγική ακρόαση. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καταλήξει σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου μία τράπεζα η οποία είτε τμηματικά ή ε, ολικά αποτυγχάνει, θα πρέπει να καταφέρει να τα βγάζει πέρα χωρίς τον φορολογούμενο. Κατά δεύτερον, ένας άλλο τομέα όπου έχει προσθεθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα έργα υποδομών, υποδομών στη μεταφορά και στις μεταφορές γενικότερα και στη μεταφορά δεδομένων. Τρίτον, στην έρευνα και την ανάπτυξη. 3% του ΑΕΠ αναλογεί στον τομέα αυτό. Αλλά θέλουμε να εξετάσουμε και το συγκεκριμένο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τέταρτον, θα πρέπει να κοιτάζουμε τις μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα, να μην αποβεί εις βάρος ε, προς τις πιστοτικές ε, διευκολύνσεις και δυνατότητες που παρέχονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρω ότι μέσω των ε, ευρωπαϊκών και των εθνικών προγραμμάτων ε, υποστηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο Βέλγιο όμως δεν φτάνει αρκετή ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται περιφερειακά, περιφερειακά προγράμματα. Αυτά κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του Βουλγικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Κλάιν από την Πολωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μυρό, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει η τράπεζά του και που συνεχίζει να πράττει στην Πολωνία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζουμε και στο μέλλον η τράπεζα να συνεχίσει να συμβάλλει αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμα σε ό,τι στην επίλυση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών προβλημάτων της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι. Η, το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συζήτηση αυτό, αυτή ε, καταδεικνύει την ανησυχία μας για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις η κατάσταση καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη και στα οικονομικά και στα θέματα προϋπολογισμού, αλλά και σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυξάνεται η ανεργία. Δεν υπάρχει αίσθηση της κοινωνικής ασφάλειας. Ο κόσμος απογοητεύεται όλο και πιο πολύ και αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωση όλο και πιο ριζοσπαστικών θέσεων και σε περαιτέρω κρίσεις, πολιτικές ε, κρίσεις, ε, ενεργειακές κρίσεις, ε, κρίσεις σε ό,τι αφορά την τιμή των τροφίμων. Όλες αυτές οι κρίσεις ζητούν και προαπαιτούν μία σωστή και δέουσα αντιμετώπιση. Ως τώρα η δράση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι πραγματικά α, οι κατάλληλε σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Γιατί τα πολιτικά συμφέροντα υπερισχύουν της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και η πρόσφατη ιστορία μας καταδεικνύει ότι ακόμα και τα μέλη της ε, ομάδας ελίτ του ευρώ, της ευρωζώνης. Δεν είναι άτρωτα. Και πάντα υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις, η ΕΠΑ, η Κίνα. Θα πρέπει πραγματικά να διαπιστώσουμε ότι η Ευρώπη ε, μένει πίσω όλο και πιο πολύ. Επικρατεί Μεγάλο σκεπτικισμός ο οποίος εκφράζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ασφαλώς διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές οι θέσεις αυτές δεν είναι δικαιολογημένες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστικοί, ρεαλιστές ε, από πολιτικής άποψης και να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Δυστυχώς, ακόμα και μια πολύ καλή διάγνωση, διάγνωση δεν επαρκεί χωρίς πράξεις, χωρίς να υπονομεύσουμε το έργο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων θα πρέπει να δηλώσουμε ότι η αντίδραση στην κρίση δεν ήταν ιδέουσα και δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική. Και φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων προβαίνουν σε όλο και πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις και το τίμημα θα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζουμε άλλη μια σημαντική απειλή η εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 θα μας φαίνεται δικαιολογημένο να ρωτήσουμε και να ρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να χρηματοδοτήσουμε την μελλοντική ανάπτυξη, αλλά τι χρησιμεύουν όλα αυτά τα μέτρα αν δεν έχουμε τα κατάλληλα κονδύλια. Πρέπει φυσικά να υπάρχει ο σχετικός προϋπολογισμός για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και αν περιορίσουμε τις, τα κονδύλια αυτά, οι στόχοι τη στρατηγικής ε, για το 2020 δεν θα είναι πολύ απλά ρεαλιστικοί. Είναι καθήκον των ευρωπαϊκών και των εθνικών ε, κοινοβουλίων να πείσουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις ότι το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Ζώνης, Ευρωζώνης εξαρτάται από την αλληλεγγύη. Θα πρέπει να βλενθούν οι διαφορέ ω προ την ανάπτυξη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το τρένο με τα 27 βαγόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ολοκληρώσει επιτυχώς το ταξίδι του. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Ιβάνοβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει δύο λεπτά στην διάθεσή της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να πούμε ότι η κοινή δουλειά μας στην Επιτροπή Κρίση, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, ξεκίνησε εδώ και 1,5 χρόνο εξετάζοντα τα αίτια και τα συνέπεια τη κρίσεως και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ήταν στοιχείο σημαντικό τη βιώσιμη ανταπόκριση στην κρίση. Η τελική έκθεση τη ομάδα αυτή για την κρίση θα κάνει συγκεκριμένε συστάσει στην πολιτική προ αυτή την κατεύθυνση και θα προσθέσει το συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα στρατηγικό όραμα για την οικονομική μα ανάπτυξη. Η διάδοση τη κρίση στην Ευρώπη επιταχύνθηκε ουσιαστικά λόγω τη ελλείψεω στέρεων δομών όσον αφορά την κυβέρνηση των φορέων και μεγάλα επίπεδα χρεών των κρατών έλλειψη επαρκών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά το θετικό τομέα. Τα σημαντικά επίπεδα των ελλημάτων και των χρεών του δημόσιου τομέα δεν μπορούν μια νυχτή να εξαλειφθούν και να μειωθούν. Αυτό χρειάζεται σοβαρά μέτρα και ισχυρό οικονομικό συντονισμό. Αυτέ οι περικοπέ δεν είναι οι λύσει αυτέ καθεαυτέ, αλλά είναι ένα απαραίτητο βήμα τόσο να εξασφαλίσουμε χρηματοστατική σταθερότητα, αν τη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο προ του στρατηγικού στόχου μα, του μακροπρόθεσμου που θα επιφέρουν την προστιθέμενη αξία στα 27 κράτη-μέλη. Έχουμε την κοινή στατική τη Ευρωπαϊκή Ενώσης του 2020 για ανάπτυξη χθε απασχόληση. Κάτι που χρειαζόμαστε, ένα καλό στρατηγικό όραμα για μακροπρόθεσμε επενδύσει. Συμφωνώ με τον κύριο Μύροφ ότι η πραγματική οικονομία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα προσέφετα ότι οι προσπάθειέ μα θα έπρεπε να εστιαστούν επί τη αυξήσεω τη ανταγωνιστικότητα τη ενώσεω μέσω συμπληρώσεω τη ενιαία αγορά και ε, να χρησιμοποιηθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει λέγαμε πάντοτε, ότι είναι στο επίκεντρο τη ενιαία αγορά Ευρώπη. Όμω σήμερα, το 2011, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μια διευκόλυνση τη πρόσβασή του στη χρηματοδότηση, κυρίω για την έρευνα και την καινοτομία και θα πρέπει να μειωθεί και το διοικητικό άχθο. Και εφόσον αναφέρθηκε η Ανατολική Ευρώπη, θα ήθελα να πω ότι σαν νέο κράτο μέλο, ανήκω σε ένα νέο κράτο μέλο και πιστεύω τα κάτι μέλη που δεν είναι στην Ευρωζώνη, θα έπρεπε να έχουν τι ίσε ευκαιρίε και να είναι σε ισότιμη βάση με τα κάτι μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ για να κανονίσουμε ποιο θα είναι, ποιε θα είναι οι προτεραιότητε στο μέλλον. Είμαστε στο ίδιο σκάφο και θα πρέπει να κολυμπήσουμε όλοι μαζί του, ώστε η προστιθέμενη αξία να υπάρχει εκεί και να δίνεται στον κάθε πολίτη. Και περνάμε στην Βουλγαρία, ο κύριος Τζόμπεφ από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα προς επίλυση. Το πρώτο είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ίσως είναι και σημαντικότερο, το σημαντικότερο θέμα. Και το δεύτερο βέβαια είναι η υποστήριξη της οικονομίας, εφόσον αυτή και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγήσουν σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έτσι θα πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης για το 2020. Όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα, βασικό μας πρόβλημα είναι το υπερβολικό χρέος. Πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει προσεκτικά με την αναγκαία μέρημνα. Πιστεύω ότι μπορούν να τα καταφέρουν οι χώρες, η χώρα μου η Βουλγαρία είχε διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα για το 2010 αλλά πάγωσε και το 2011 μόνο το έλλειμμά μας ήταν μόλις 2,5% του προπολογισμού δηλαδή 2,5% και εξετάζουμε ένα σύμφωνο ανάπτυξη αθερότητας για τη Βουλγαρία εκεί θα πρέπει ο δημόσιος τομέας να συμμετέχει δεν θα πρέπει να ξεπερνά ο δημόσιος τομέας το 97% του ΑΕΠ δεύτερον το έλλειμμα του προπολογισμού θα πρέπει να είναι ευέλικτο και κάτω 3% και θα πρέπει να καθορίζεται από την οικονομική ανάπτυξη και από την ύφεση, ανάλογα με τον κύκλο. Πάνω κάτω, εντός όμως του ορίου του 3%. Τρίτον θέμα είναι η φορολογική πολιτική. Πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής, δεν θα πρέπει να αλλάζει κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί έτσι μια βιώσιμη ανάπτυξη και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Προβλέπουμε ότι θα αλλάξει το φορολογικό πλαίσιο στη Βουλγαρία αν το αποδεχτούν τα δύο τρίπτα των μελών της Εθνοσυνελεύσεως. Θα δημιουργηθεί έτσι εξοπιστία για τους επενδυτές και δημιουργηθεί το αναγκαίο περιβάλλον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δημιουργηθεί απασχόληση. Επιτυγχάνοντας λοιπόν την οικονομική σταθερότητα και στηρίζοντας την οικονομία στο σύνολό της και πιο συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φρονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να πετύχει μακροπρόθεσμες επενδύσεις για ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Καλό τώρα τον Λούρο Ζεύσικ από την Τσεχική ε, Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι μετά από δέκα χρόνια που εξασκώ τα καθήκοντά μου έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ε, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελάχιστος βρήκα που να είναι ε, τόσο έμπειροι όσο η αντιπροσωπεία της οποίας ηγούνται ο κύριος Κλίντς και ο κύριος Κάρας και ε, γι' αυτό θα έπρεπε να βρούμε ε, μία λύση στο ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστώ για τη δημοσίευση του εγγράφου. Ξέρω ότι έχετε επισκεφθεί πολλά κοινοβούλια και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε αυτές τις επισκέψεις. Σε μία από αυτές τις πράξεις βλέπουμε ε, την γέφυρα του Καρόλου, ένα μνημείο της χώρας μου όπου έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένες περιπτώσεις όπου η γέφυρα αυτά μετά από φυσικές καταστροφές, μετά από πλημμύρες έσπασε, χρειάστηκε αριθμό ετών για για να μπορέσει να επιδιορθωθεί και ελπίζω ότι ε, οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο θα αντιπεξέλθουν των κρίσεων που έχουμε, ε, αντιμετωπίσει και στο παρελθόν χάρη στην εργασία, χάρη στις μεταφράσεις έχετε όλη τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την θέση του, της γερουσίας της Τσεχίας και ήθελα να σας πω ότι θα μιλήσουμε συχνά για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μια εξέχουσα αξία. Είναι απαραίτητη τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν ελλείψεις αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω δεν πρέπει αυτή η αλληλεγγύη που είναι ευγενές, ε, ε, ευγενής αρχή ε, με τα πηδήσουν εις μία υπερβολή που θα είναι εις Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Φιλανδίας, ο κύριος Σάριος. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Κρίσεως και πρέπει να σας πω ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Διότι ε, είχαμε την ε, διάσκεψη κορυφής το Σαββατοκύριακο όπου ε, συζητήσαμε για το ρόλο της Πορτογαλίας η οποία δραστηριοποιήθηκε ε, η χώρα αυτή ε, έβαλε αμέσως μέτρα και δεν επεκτάθηκε σε αυτήν η κρίση και εδώ συνδυάζω το σχόλιο μου με αυτά που είπε ο κύριος Κύρο δηλαδή θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να βρίσκεται στο προσκήνιο η οικονομία και ε, να δούμε ε, πώς θα αντεπεξέλθουμε και πρέπει να δούμε τι μαθήματα έχουμε αποκομίσει από την κρίση. Βλέπουμε ότι οι τράπεζες θα υποβληθούν σε ένα νέο stress test και θα πρέπει αυτό να είναι πιο αποτελεσματικό αλλά γενικώ η Ευρώπη δεν έχει καμία δυνατότητα να αντεπεξέλθει αυτού του stress test όταν απλώς γίνεται σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα σημεία από τα οποία δεν έχουμε διδαχθεί όπως είπαν και προλαλήσαντες διότι οι τράπεζες λαμβάνουν ακόμη λανθασμένες αποφάσεις και ε, οι αποφάσεις αυτές συνεχίζουν παρόλο που ξέρουμε ότι ήταν λαθασμένες οι αποφάσεις αυτές άρα η κατάσταση δεν μας δίδαξε τίποτα. Ε, πρέπει να υπάρχει μια κοινή ενέργεια. Ε, βλέπω εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου μου και το πρόβλημα μου τώρα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη λύση. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ο ευρωσκεπτικισμός αριθμός αυξάνεται συνέχεια και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διαβλέπω τον κίνδυνο να ε, αντιμετωπίσει προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει τα θέματα που μας απασχολούν. Ε, υπάρχει ένα θέμα όπου οι εθνικοί βουλευτές έχουν ε, ιδιαίτερη ευθύνη πρέπει ε, να αντιληφθούν ε, οι πολίτες κάθε χώρα στη σημασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το 2020. Υπάρχει, ε, υπάρχουν θετικές απαντήσεις ή το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Κρίσεως, ιδίως αν δούμε το θέμα του, της φορολογίας των χρηματοοικονομικών κινήσεων Βλέπουμε ότι προβλέπεται για τις συναλλαγές ε, μια φορολογία την οποία έχει προωθήσει δις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της εκθέσεως της Άνης Ποδηματά στο Στρασβούργο και ε, έχω ακόμη δύο λόγια μόνο να σας πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει και ίδιου πόρους. Αυτή είναι καλή ιδέα και ε, ελπίζω θα έχει και καλή έκβαση. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ και τώρα καλό τον κύριο Μάτς Νιτέρ από το Αυστριακό Κοινοβούλιο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε πολύ σαφώς ο κύριος Μύρο. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο ε, ε, φτάσαμε σε καινούργια μεγέθη και χρειαζόμαστε πραγματικές επενδύσεις για να υπάρξει παραγωγή αλλά αυτό δεν γίνεται και αυτό δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύο-τριών ετών αλλά πολλών δεκαετιών. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε γιατί αν δεν το λύσουμε η βιώσιμη Ευρώπη δεν θα αναπτύσσεται. Όπως όσο έχει ε, αναπτυχθεί ανεπαρκώς στη δυτική πλευρά επί τα τελευταία 15-20 χρόνια γιατί έχουμε ένα πρόβλημα χρεών το οποίο δεν έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πρότυπο της, ε, της ε, ε, Ευρώπης για την ανάπτυξη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω χρηματοδοτήσεως από τις τράπεζες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ δεν πρέπει να συζητάμε μόνο για το πώς θα ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές αλλά ιδίως πώς θα βρούμε χρηματοδότηση. Γι' αυτό και χαιρετίζω το πρότυπο, πρότυπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διότι πρέπει να δούμε αν δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις τράπεζες με νέους θεσμούς. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στο βελγικό, στη βελγική γενουσία και δίνω το λόγο στον κύριο Λαουέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε συμφωνώ με αυτά που είπε ο αυστριακό ε, συνάδελφο, να υπενθυμίσω ένα στοιχείο εκθέσεως οικονομολόγου που επιδόθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που υπενθυμίζει ότι οι χρηματοστικέ συναλλαγέ ε, είναι 3, ε, δολάρια το χρόνο σαν τζίρο. Και μετά από μελέτη της, του Πανεπιστημίου τη Τουλούζη, η παροχή υπηρεσιών, η, η επίδοση αγαθών, η πραγματική οικονομία δηλαδή, είναι μόλις το 2% αυτών των 3-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή προσπάθειες που κάναμε μέχρι τώρα για να ρυθμίσουμε με καλύτερο τρόπο τα χρηματοστατικά δεν νομίζω ότι μπορούν να απορροφήσουν αυτή τη φυσαλίδα. Χωρίς την απορρόφηση αυτή δεν μπορούμε να ξαναδώσουμε στην πραγματική οικονομία την πραγματική της θέση που της ανήκει. Δηλαδή ε, να έχει πραγματική θέση στα χρηματοστατικά, τα οποία χρηματοστατικά πρέπει να είναι τα μέσα και όχι να επικρατούν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και ανησυχώ περισσότερο ακόμα βλέποντας τις εργασίες της Βασιλείας Τρία που αντικειμενικά πιστεύω ότι οι δραστηριότητες εκτός προπολογισμού τραπεζικού τομέα δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα που θα πρέπει να το καλύψουμε. Τρίτο στοιχείο της παρέμβασής μου με το οποίο θα κλείσω. Δεν θα ήθελα εδώ ε, να τοποθετηθώ μεταξύ οικονομίας της προσφοράς και οικονομίας της ζήτησης. Απλώς παρατηρώ ότι εδώ και 30 χρόνια περίπου η κατάσταση των εργαζομένων όσον αφορά την οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Κατά 10% όσον αφορά, η μισθή όσον αφορά ποσοστό το ΕΠ έχει υποχωρήσει κατά 10%. Και δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χωρίς να έχουμε εργαζομένους οι οποίοι απολαμβάνουν επίπεδο διαβίωσης επαρκές για να μπορέσουν να βασιστούμε επ' αυτής μια οικονομία της ζήτησης και εκεί να βασίσουμε την ανάπτυξη και όχι στην ανταγωνιστικό των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή καλύτερη του πλούτου και η οποία θα πρέπει να οδηγήσει στο να καλύψουν το χαμένο έδαφος οι εργαζόμενοι. Ο Λεϊσμίτα από τους Φιλελεύθερους, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλή σωστό το ότι αναφέρατε την Ιαπωνία. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες ε, εκτιμήσεις για το πώς πρόκειται αυτό να επηρεάσει την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη και το πώς ε, αντιδρούμε στην ε, κρίση του κλίματος. Επίσης, χάρηκα που αναφερθήκατε στην Βόρεια Αφρική, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία για εμάς στην Ευρώπη, αντί να φροντίσουμε τους μετανάστες. Φυσικά και πρέπει να αναλάβουμε τις Ευθύνε μας, αλλά καλύτερα θα ήταν να αγοράζουμε τα προϊόντα τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εδώ στο Κοινοβούλιο τα βασικά σημεία της πολιτικής μας. Επίσης, ε, να αναφερθώ σε αυτό που ανέφερε και η συνάδελφος Ιβάνοβα σε ό,τι αφορά το ευρώ και το σύμφωνο για το ευρώ. Με απασχολεί αυτό ιδιαίτερα, αν και προέρχομαι από μια χώρα εκτός της Ευρωζώνης, η Βελγική Προεδρία ε, και εδώ ο Βέλγος εκπρόσωπος ήταν πολύ ικανοποιημένος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος για κάποια από τα συμπεράσματα, αλλά ανησυχώ ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι αυτό θα ε, οδηγήσει σε μια Ευρώπη δυτή. Οι χώρες ε, της Ευρωζώνης θα κινούνται με μια αλφα ταχύτητα και τα υπολείμματα οι υπόλοιποι θα ξεμείνουν. Και τελικά το συμπέρασμα θα είναι ότι θα αποφασίσουν πράγματα τα οποία θα καλούμαστε εμείς απλά να αποτεχτούμε εκ των υστέρων. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε και θεωρώ αυτό ότι θα ήταν επιζήμιο, όχι όμως πολιτικός, αλλά και για τη βιωσιμότητα της ενιαίας αγοράς και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ένα από τα ευρωπαϊκά είδωλα, τον κύριο Ντελόρ, σήμερα το βράδυ στο δείπνο να μας εξηγήσει τι θεωρεί ότι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα και τι γίνεται με την κοινωτική μέθοδο, η οποία δεν θεωρώ ότι έχει πετύχει να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Ευχαριστώ και τώρα εκπρόσωπος του Bundesrat, ο κύριος Μάρκοφ από τη Γερμανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να πω ότι ως Υπουργός Οικονομικών του κρατηδίου του Μπραντενμπουργκ ε, έχω απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ότι για το ψήφισμα του 20 Οκτωβρίου του 2010 θεωρώ ότι απεικονίζει και εξηγεί πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Τα διάφορα θέματα 7, 19, 47, 121, 151, 158 και 219. Όλα αυτά τα σημεία μπορείτε να τα διαβάζετε μετά. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Επίσης, να συμφωνήσω με κάποιους συναδέλφους. Νομίζω ότι κάποια προβλήματα δεν έχουν αναφερθεί, γιατί εξακολουθούν να αυξάνονται τα ε, ρευστότητα των πλενασμάτων και δεν έχουν λυθεί πολλά ζήματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι τράπεζες οι τράπεζες δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία γιατί είναι πολύ περιορισμένα τα επιτόκια. Θα συνεχίσουν να πουλάνε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθεσία. Αυτά σε προσπάθειες αυτορύθμισης δεν πρόκειται να πετύχουν όπως δεν πέτυχαν και στο παρελθόν άλλωστε. Το επόμενο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι στη συζήτηση θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι διαφορετικές ε, ε περιφερειακές ε, καταστάσεις και συνθήκες. Στο Βραντεμβούργο, για παράδειγμα, δεν έχουμε εξαγωγές, είμαστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να εξέλθουμε τις κρίσεις. Όλες αυτές οι διαφορές πραγματικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα διάφορα μέσα τα οποία θα προταθούν. Τελευταία παρατήρηση. Ε, μας στείλετε και ένα ερωτηματολόγιο σε ό,τι αφορά την ε, επενδυτική πολιτική. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν επενδύσεις μετακύλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιοριστούν τα χρέη και το τελευταίο σημείο γρήγορα γρήγορα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί ένα νέο σύστημα νομοθεσίας ε, παρέμβασης. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Να μην, ε, να μην επιτρέπουμε σε μικρές επιχειρήσεις να προβάνουν σε πτώχευση, αλλά τώρα η κυρία Παπανδρέου, λέει ο, κύριος, ο πρόεδρος από την Ελλάδα. Το μικρόφωνο σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο για την ε, παρουσίαση και πράγματι νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η Sustainable Growth Model. Συμφωνώ ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία να ξανακαθορίσουμε τον ε, τομέα το χρηματοπιστωτικό και η οικονομία να γίνει πιο πράσινη. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά όταν μετά από δύο χρόνια από την ε, κρίση στην οποία βρισκόμαστε και νομίζω σε αυτό το σημείο υπάρχει γενική συμφωνία ότι ο κύριος λόγος ήταν ο τρόπος λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα βήματα που έχουν γίνει προς τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για πιο αποτελεσματικό έλεγχο είναι πάρα πολύ ε, μικρά και αντίθετα βλέπουμε ότι το χρηματοπιστωτικό τομέας ε, κατάφερε το 2010 να έχει πρωτοφανή κέρδη. Ε, πώς μπορεί να συνδυαστεί η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με το πακέτο αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που βεβαίως πρέπει να ελέγξουμε τα, τα ελλείμματα και το χρέος αλλά πώς είναι δυνατόν να μειώνουν όλες οι χώρες ή να υποχρεούνται να μειώσουν, δεν μιλάω για την Ελλάδα που είναι μια ειδική περίπτωση, μιλάω για όλες τις χώρες στην Ευρώπη, τις δαπάνες για στην παιδεία, στην ε, ε, εκπαίδευση, στην ε, υγεία, αλλά και στις επενδύσεις στα infrastructure και ποια είναι η δική μας ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Χρειαζόμαστε, είπατε, ένα well-educated workforce. όταν όμως μειώνουμε αυτές τις δυνατότητες, δεν υπονομεύουμε τις προσπάθειες ε, της Ευρώπης στο μέλλον. Μήπως με τις πολιτικές οι οποίες είναι one-sided ε, θα δημιουργήσουμε μια γενιά, ε, χαμένη γενιά. Εγώ θα συμφωνήσω με τη συζήτηση που γίνεται για την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι όμως δυνατόν να υπάρχουν το ίδιο μοντέλο, το γερμανικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, να υποχρεωθούν όλες οι χώρες να το εφαρμόσουν. Είναι δυνατόν οι άλλες χώρες να εφαρμόσουν ένα μοντέλο που είναι λίγο ξεκομμένο από την οικονομική, την κοινωνικό, κοινωνική τους κατάσταση. Δηλαδή, τελειώνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ τον ε, κύριο Φεώτη από την ε, Πορτογαλία να Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι Ευρωβουλευτής από την Πορτογαλία. Είμαι μέλος Επιτροπής ΚΡΙΣ και στο δίλεπτό μου θα ήθελα να εκφράσω μία-δύο ιδέες. Καταρχάς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση με μέτρα λιτότητας. Στη χώρα μου αυτή τη στιγμή, στην Πορτογαλία, συζητούμε τα μέτρα λιτότητας. Αλλά δεν αναφέρονται οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις, όλος ιδιαίτερος μεταρρυθμίσεις του επενδυτικού τομέα, μεταρρυθμίσεις στην αγορά, στην αγορά εργασίας, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική πολιτική όσον αφορά το χρηματοστητικό σύστημα για τις χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να ταιριάζει σταθερότητα με την ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε και σε εθνικό επίπεδο μέτρα. Να βρούμε σε εθνικό επίπεδο επίσης ε, λύσεις. Παράλληλα με την ευρωπαϊκή λύση. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την οικονομική διακυβέρνηση και ας χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ούτω ώστε να έχουμε τελικά μια ενιαία πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει σε αντιμετώπιση της κρίσης. Το σύμφωνο για, τις, το ευρώ ίσως να έχει θετικά αποτελέσματα, ίσως να αποτελέσει έναν μηχανισμό που θα μας οδηγήσει σε επίλωση, επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου και ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Θέλουμε μια Ευρώπη που να κινείται όλοι με μια ταχύτητα. Θέλουμε περισσότερη ε, ολοκλήρωση, περισσότερη αλληλεγγύη, κοινό όραμα, περισσότερη Ευρώπη. Και σχετικά με αυτό πρέπει να πω ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι κρισίμου σημασία που συζητούν με πολύτιμο τρόπο την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ζων Ρομπέρ από την ε, Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν αναφέρατε την στρατηγική της Λισαβόνας και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να σημειώσουμε αυτή την αποτυχία αλλά η δουλειά που πρέπει ε, να κάνουμε τώρα δεν πρέπει να είναι εις βάρος των συμπολιτών μας οι οποίοι δεν θα πιστεύουν πλέον ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους. Θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω πει επανειλημμένο σχετικά με το χρέος ότι στην τελευταία περίοδο η γενιά μας κατάφερε ότι δεν μπορεί να μην πληρώσει αυτό το χρέος και να το μετακυλήσει στα παιδιά της. Αλλά ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να επαναλάβουμε είναι ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες και έτσι να ξεπληρώσουμε το χρέος διότι έτσι μειώνουμε έχουμε τις ε, δαπάνες συνοχής υγείας, παιδείας, ε, μελλοντικών επενδύσεων ε, τις οποίες χρειαζόμαστε. Πώς θα λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα Αντί για νέα φορολογία θα πρέπει να υπάρχει ε, άλλη μορφή φορολογίας το οποίο να αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας όπως και σε άλλες. Υπάρχει η νέα ανάπτυξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πράσινη ενέργεια, όλα αυτά τα επιθυμούμε. Αλλά πώς θα τα επιτύχουμε και αν θα ε, χρηματοδοτήσουμε μέσω ενός συστήματος ευρωπαϊκού δανείου δεν θα πρέπει να υποκαστήσουμε στη, στα χρέη των ε, κρατών μας ένα χρέος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί έτσι δεν θα έχουμε αλλάξει τίποτα και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η φορολογία των χρηματοοικονομικών πράξεων ε, που είναι πολύ αμφιλεγόμενο και τέλος οι τράπεζες δεν μπορούμε να προσβλέπουμε στο μέλλον χωρίς να ενδιαφερθούμε εις ε, τις παρεκκλήσεις του τραπεζικού συστήματος ε, όπου συμφωνώ ότι δεν έχουν λυθεί και αυτό που μας προτείνεται μέχρι στιγμής δεν θα τις λύσει. Ευχαριστώ και δίνω τώρα το λόγο στον Τζαν Κάρλο Ζοζέτη. Απουσιάζει. Λοιπόν, θα έρθει αργότερα. Τότε την Ελίζα Φερέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κρίση αυτή έριξε πολύ φως στην Ευρώπη. Έδειξε ότι η Ευρώπη έχει πολύ μειωμένα μέσα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κρίσεις δεν έχουμε μέσο μακροπρόθεσμο όραμα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε και όχι να αντιδρούμε. Ο διακυβερνητικός χαρακτήρας, διακυβερνητική προσέγγιση ενισχύθηκε τελικά από την κρίση. Η κοινοτική μέθοδος ε, έχασε έδαφος. Πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Η Ευρώπη σημείωσε κάποια πρόοδο, κυρίως όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι καλές συνθήκες αυτές, αλλά δεν αρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό που συμβαίνει τώρα, στην κρίση του ευρώ, μας δείχνει κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η χρηματοπιστωτική κρίση έγινε μια κρίση της πραγματικής οικονομίας, μετά έγινε κοινωνική κρίση και γίνεται και κρίση εθνικού χρέους. Και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αυτή η, αυτή η κρίση να ξεχυλήσει και να επηρεάσει και την πολιτική ζωή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα ήταν θανατηφόρο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν έχουμε πρόβλημα όπως έχει το δολάριο. Ε, έχουμε όμως διτό πρόβλημα όσον αφορά το ευρώ. Λοιπόν, ποιος είναι ο χαρακτήρας του προβλήματος, ο διτός. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξή μας είναι ανεπαρκής σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ οικονομιών της Ευρωζώνης και αυτό επιδεινώθηκε λόγω του ότι υπάρχει μια πολιτική ενία οικονομική και εμπορική λόγω του ενός νομίσματος. Και αυτό αναφέρθηκε σε σχετική έκθεση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή και Νοσματική Ένωση. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν τώρα βασικά είναι να επιστρέψουμε στο παλιό πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής, ούτω ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μια πραγματική σύγκληση, σύγκληση παραγωγικότητας ημερομισθείων και άλλων συνιστοσών της οικονομίας. Θα πρέπει το σύμφωνο το σύμφωνο ανταγωνιστικότητα δεν θα λειτουργεί αν το μόνο διθωτικό μέτρο που θα λάβουμε θα είναι η μείωση των αντί να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα με έναν σε ένα πλαίσιο σύγκλησης. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακροπρόθεσμα, σε μεγαλύτερο βάθος όταν εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι είδους πρόγραμμα έχει η Ευρώπη σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ούτω ώστε να μπορεί η Ευρώπη να χειριστεί την εξωτερική της πολιτική, την εμπορική της πολιτική. Ποιο είναι το πρόγραμμα στα πλαίσια του G20, τι γίνεται με τη φορολογία τι εργαλεία συνοχής έχουμε στη διάθεσή μας που είναι προσαρμοσμένα στον 21ο αιώνα και εν τέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τέτοιες διαφορές μεταξύ οικονομιών και με τόσο χαμηλό προϋπολογισμό ευρωπαϊκό. Έκανε σχετικά κάποιες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα ηγηθούμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Από τη Ρουμανία παρακαλώ τώρα εκπρόσωπος. Εκτός μικροφώνου. Μικρό, μικρό. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ψήφισμα αυτό που ανέφερε και ο κύριος Μύροφ. Συμφωνώ και είναι πολύ σημαντικά αυτά που ανέφερα. Κάποια σχόλια να κάνω το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος είναι τόσο υψηλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Μιλάμε για το κρατικό μοντέλο το οποίο προάγουμε και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλάβουμε τον κίνδυνο και να εξετάσουμε τον, επανεξετάσουμε το ρόλο που παίζει το κράτος, να δούμε ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του κοινωνικού κράτους και της κρίσης να υπολογίσουμε πόσα χρήματα χαραμίστηκαν σε επενδύσεις για δημόσιες δαπάνες, καλύπτοντας τα ελλείμματα και το κόστος του δημοσίου χρέους. Αν προβούμε σε μια τέτοια ανάλυση σε ό,τι αφορά το δημόσιο και το δυτικό χρέος, για μια χώρα, χώρα όπως η Ιταλία βλέπουμε ότι το κράτος όπως ήταν οργανωμένο τις τελευταίες δεκαετίες ήταν πιο ακριβό. Και παρά το γεγονός που ότι εξακολουθούν τα χρέη να είναι τόσο ψηλά, τα συστήματα, ιδιαίτερα το σύστημα συνταξιοδότησης, αποτυγχάνει. Ουσιαστικά τι κάνουμε, επιδεινώνουμε και αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στην ε, χρηματοοικονομική πολιτική αυξάνουμε τις δαπάνες. Και για παράδειγμα, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα αν προκαλούμε πολλά, πολλές επιπρόσθετες δαπάνες κατά τη διαδικασία της υπερβολικής ρύθμισης, της υπερβολικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τα χρηματοπιστωτικά. Κοιτώντας για παράδειγμα την τιμή του πετρελαίου σε άλλες, τιμές, σε άλλες περιοχές του κόσμου, βλέπουμε ότι δυστυχώς με, τα, με τους δασμούς αυξάνουμε το κόστος και μειώνουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Και τελευταίο σημείο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να επικεντρωθούμε πιο πολύ στην έρευνα και να δημιουργηθεί μια κοινή πολιτική στον τομέα αυτό για να γεφυρώσουμε το χάσμα με τη Βόρεια Αμερική. Για να αυξήσουμε το ρόλο της Ευρώπης, να τον τονίσουμε το ρόλο της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο σε, στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος, οι δύο τελευταίοι εμελητές από τη Λιθουανία, ο κύριος Κάιτιας και ο Τόμας Μαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το ΕΛΚ. Ο κύριος Κάιτιας πρώτος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Λιθουανία θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσης το 2013. Προσπαθούμε να μάθουμε τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και τονίστηκε από προηγούμενους ομιλητές η παραγωγή, η παραγωγικότητα. Οι τράπεζες πολλούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία προϊόντα αυτά δεν έχουν μεγάλη σχέση με την παραγωγή, ούτε με την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων έχει υποφέρει πολύ η χώρα μου από την κρίση, η Λιθουανία από την κρίση και πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα να βρει δουλειά διότι τα προσόντα τους δεν αρκούν για την αγορά εργασίας και ο κόσμος θέτει ερωτήματα. Λένε γιατί δεν κατασκευάζουμε εργοστάσια στη Λιθουανία και δημιουργούνται αμφιβολίες. Ε, υπάρχει έλλειψη περιφερειακής συνεργασίας. Ε, η ανατολική εταιρική σχέση. Ο κύριος Μύροφ αναφέρθηκε για, στη Volkswagen που θα μπει στη Ρωσία και θα μπορούσαμε και εμείς να συμμετάσχουμε σε τις αγορές. Και η ανάπτυξη λοιπόν της παραγωγής μέσω συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Αναπτύξεως θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια λύση. Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια Ευρώπη δύο και τριών ταχυτήτων. Και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, το οποίο υπογράφεται τώρα, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες. Φαίνεται σαν να χάνει έδαφος η κοινοτική μέθοδος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε περισσότερο στην κοινοτική μέθοδο για την επίλυση των προβλημάτων. Όσον αφορά το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μπορούμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι τράπεζες να στραφούν περισσότερο προς την παραγωγή, διότι χωρίς αυτό η οικονομική, ανάπτυξη δεν θα σχετιστεί με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστώ δύο λεπτά κύριε Στόμασμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να γίνουν πιο ορατές στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά συμφωνώ και με τον συνάδελφο που ανέφερε ότι υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάσταση και αυτή θα πρέπει να καταστεί ε, καλά διακριτή. Θα ήθελα να πω ότι Μύρο, έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Αντιμετωπίζουμε μια φάση δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λέξη ρεαλιστική για την επέκταση του προϋπολογισμού μας σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, το θέμα του φρένου στα χρέη, το θέμα είναι επικαιρό. Και κατά δεύτερο να μας πείτε πώς η τράπεζά σας θα συνεργαστεί και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε τέτοια χρηματοδότηση προγραμμάτων. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σχέση, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό ε, σε ό,τι αφορά τη μεταξύ σας συνεργασία και για την χρηματοδότηση σχεδίων. Έχουν να κάνουν με projects στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και κάποια ποσοστά ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για κάποια project στη Ρωσία και στην Ουκρανία και αν προβλέπετε τέτοια σχέδια. Είναι σημαντικό το θέμα της βιωσιμότητας. Υπάρχει ε, στην τράπεζά σας ένας ορισμός της βιωσιμότητας για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ο ίδιος, ε, η ίδια αντίληψη σε ό,τι αφορά όλη την Ευρώπη. Και τελευταία ερώτηση, όταν κάποια project είναι κοινή ωφελία. Θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από την τράπεζά σας ακόμα και αν είναι περιορισμένη η απόδοση η οποία αναμένεται. Υπάρχουν κάποια τέτοια κριτήρια απόδοσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και θα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μύρο και να πω ότι ο κύριος Μύρο έχει χρονικούς προορισμούς και μετά από την απάντησή του δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσει, πολύ λυπούμαστε, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ως απάντηση στις ερωτήσεις του. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και στα ενδιαφέροντα σχόλια. Δεν θα είναι αυτό δυνατόν, θα πρέπει να περιοριστώ και να κάνω τρία ή τέσσερα ε, επιπρόσθετα σχόλια. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ε, Ευρώπη, επειδή αναφέρθηκε η έννοια του ευρωσκεπτικισμού και δικαίω αντιλαμβάνομαι, θεωρώ ότι καταρχάς είναι πολιτική η φύση της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε και η πολιτική πρόκληση είναι η εξής. Πώς θα αντικαταστήσουμε τους, την νοτροπία η οποία επικρατούσε μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ένωση της Ευρώπης με μια ε, νοτροπία η οποία θα πείσει το κοινό του σήμερα και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε τα διάφορα θέματα για το τι μπορούμε και θα έπρεπε να κάνουμε ή να κάνουμε καλύτερα. Αν συνεχίσουμε να παρατηρούμε αυτά που παρατηρούμε σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ότι η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητείται, δεν θα πετύχουμε. Λοιπόν, ζητώ κατεπηγόντως πολιτική ηγεσία. Να βγούμε και να διατρανώσουμε ότι αν η Ευρώπη δεν συνεχίσει ενωμένη σήμερα θα χάσουμε οποιαδήποτε σημασία σε οικονομικούς όρους και σε ό,τι αφορά την ε, τις αξίες μας σε όλο τον κόσμο. Δεύτερη παρατήρηση για θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα. Φυσικά, πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι το να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μικρών δυναμικών, το να συνεχίσουμε να ρυθμίζουμε τις τράπεζες, να αυξήσουμε τις κεφαλογικές για τους μεμονωμένους φορείς, αλλά τελικά να μην καταφέρουμε να ελέγξουμε τις αγορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αγορές over the counter και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που δεν υποκίνται σε ρυθμίση και σε ένα βαθμό που θα συνεχίσει να διευκολύνει τους φορείς αυτούς και τελικά τον κίνδυνο να τον αναλαμβάνει ο φορολογούμενος. Δεν θα καταφέρουμε να διοχετεύσουμε τις επενδύσεις στους τομείς που επιθυμούμε να διοχετευτούν. Τρίτη παρατήρηση. Για θέματα δημοσίου χρέους και λιτότητας. Καταλαβαίνω όσους ισχυρίζονται ότι η χώρα τους αντιμετωπίζει δυσκολίες να ακολουθήσει τέτοιες ε, μεθόδους εις βάρος των μελλοντικών γενεών. Τι εναλλακτική έχουμε όμως, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα συστήματα με τρόπο που θα είναι αποδεκτό από τις αγορές, γιατί κάθε χώρα, κάθε οντότητα πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να αντέχουμε το επίπεδο των χρεών που έχουμε σήμερα, χωρίς να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα χρειαστούν τα χρήματα του φορολογούμενου για την κάλυψη των επιτοκίων αντί για την επένδυση σε δημόσια αγαθά. Όσο δύσκολο και να είναι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να ομολογήσουμε ότι έχουμε μαζέψει πολλά αναποτελεσματικά συστήματα και αυτά τα συστήματα τα αναποτελεσματικά έχουν οδηγήσει με τη σειρά τους σε πολλές περιπτώσεις σε μεγάλη συμμετοχή δημοσίου χρέους και τα δημόσια χρέη πλέον αυτά είναι μη βιώσιμα. Ως εκ τούτου, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαιρεθεί, θα γλιτώσει. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι τμήμα των χωρών εκείνων που θα πρέπει να αναλάβουν, να λάβουν μέτρα λιτότητας. Έγινε ένα σχολείο για την ενέργεια σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία. Και προφανώς χρειάζεται προσοχή εν ώψη και όσων συμβαίνουν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Ένα όμως είναι απόλυτα σίγουρο. Οι επενδυτές στον κλάδο αυτό χρειάζονται ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο και αυτό που πραγματικά ε, χαλάει την κατάσταση στην παρούσα φάση και το ακούω αυτό λιμερής από τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τις επιχειρήσεις του οικονομικού κλάδου που σκέφτονται να επενδύσουν. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν ξέρουν αν αυτά που ισχύουν σήμερα θα εξακολουθούν να έχουν αξία αύριο. Και όσο δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με για μια ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ενέργεια δεν θα καταφέρουμε να δώσουμε κίνητρο για τις επενδύσεις και ξέρω πάρα πολλές επενδύσεις, πολλές εταιρείε που έχουν πάρα πολλά χρήματα αλλά δεν τα επενδύουν γιατί, γιατί, γιατί έχουν ένα επιχείρημα. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στο νομικό πλαίσιο το οποίο στην παρούσα φάση υπάρχει. Άρα απευθύνω κατεπίγουσα έκκληση. Ακόμα και αν χρειαστούν συμβιβασμοί, σας καλώ να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις ενεργειακές επενδύσεις το οποίο θα κρατήσει πέρα από ένα χρόνο και πέρα από μια πολιτική πλειοψηφία για τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, κύριε Μαν, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να το συζητήσουμε διάν γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σας. Όπως είπα όμως, θεωρώ, και τώρα δεν σας μιλώ ως ε, πρόεδρος μιας τράπεζας, αλλά ως άτομο το οποίο δεσμεύεται πλήρως για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας μιλώ και σας λέω ότι θεωρώ ότι όλες οι καλές συμβολές, όλες οι καλές συστάσεις, όλα τα καλά συμπεράσματα τα οποία θα εξαγάγετε από τις συζητήσει σας, για τις οποίες πραγματικά τρέφω μεγάλο σεβασμό, θα οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα μόνο, μόνο εφόσον υπάρχουν οι πολιτικοί όροι. Και οι βασικοί πολιτικοί όροι είναι οι εξής. Να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Uh, Δυστυχώ θα πρέπει να φύγει ο κύριο Μύρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μα και την πρόσκλησή μα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σα. Εμεί συνεχίζουμε. Και τώρα έχουμε ένα γύρο συντονιστών από τις πολιτικές ομάδες. Δύο λεπτά ο καθένας. Πρωτού ωστόσο σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μία συνάδελφο από την Πορτογαλία, στην κυρία Μάρτινς, η οποία ζήτησε το λόγο, αλλά σας δίνω μόνο ένα λεπτό. Μα πού είσαστε? Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για τη χώρα μου. Πρόσφατα, σημαντικές επενδύσεις εστιάστηκαν επί βασικών τομέων, δύο βασικών τομέων, επί της παιδείας και επί της ερευνάς. Κάναμε και διάφορες διαθωτικές μεταρρυθμίσεις στην Πορτογαλία. Αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές, όπως η σημερινή, και είναι καλό η Επιτροπή αυτή που Επιτροπή ταξίδευσε στην Πορτογαλία και ήρθε σε επαφή με διάφορους βουλευτές για να ακούσει απόψεις. Όπως έλεγα όμως παρά τις εφαρμοστήσεις μεταρρυθμίσεις, παρά τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθώ να πιστεύω ότι πολλές χώρες, πολλοί κόσμος στην Ευρώπη δεν εγνώριζαν ότι έγιναν διαθωτικές αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και στην Πορτογαλία μάλιστα. Θα πρέπει να εστιαστούμε, όπως είπατε, πράγματι επί της πραγματικής οικονομίας. Και θα πρέπει οι τράπεζες και η οικονομική πολιτική να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία και όχι το αντίστροφο. Συμφωνώ με τους δύο συμπατριώτες μου που μίλησαν προηγουμένως και αναφέρθηκαν στο θέμα. Στην Πορτογαλία και εμείς στην Ευρώπη συζητούμε άλλα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Αν είχαμε πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Καμιά φορά εστιαζόμαστε αποκλειστικά στα ελλείμματα. Νομίζω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά το θέμα των δαπανών και της μειώσεως των δαπανών, διότι αυτό είναι κάτι που ήδη επηρεάσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα παίρνουν το λόγο οι συντονιστές και καταρχήν ε, ο κύριος Έγγελ για το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον κύριο Μυρό, με αυτά που μας είπε. Είπε ούτε, ότι είτε θα καταφέρει να κάνει τη δουλειά της ολοκλήρωσης η ε, Ευρώπη. Αλλιώς θα χάσει τη θέση στην ε, παγκοσμιοποιημένη υφήλιο. Αυτό είναι το θέμα. Όσον αφορά τη συζήτηση, τέσσερα συμπεράσματα έχω συναγάγει. Συζητήθηκε η αγορά. Είναι θέμα αυτό και αναζωγόνηση αυτής. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξή. Όλα αυτά στρέφονται γύρω από την αναζωγόνηση μιας οδηγίας που τον παλιό καλό καιρό θα έπρεπε να έχει το όνομα του συντάκτου του, του Φρίτς Μπόλκενστάιν. Μπορούμε να επιμείνουμε επί όλων των προόδων που προτείνει και ο καθηγητής Μόντι, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει πιθανότατα θα πρέπει ε, να γίνουν φιλελευθεροποίησεις που δεν βρίσκουν όλη την Ήπειρο ε, σύμφωνη. Δεύτερον, ανάπτυξη και τι γίνεται το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Εν πρώτης, η Ευρώπη πιθανότατα θα πρέπει να διαπιστώσει ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε πλέον την παλιά γνωστή ανάπτυξη, τουλάχιστον παντού, και δεν θα συγκρίνεται με αυτά με την ανάπτυξη άλλα μέρη του κόσμου. Και πάνω απ' όλα δεν μπορούμε να αγοράζουμε συνεχώς ανάπτυξη. Είδαμε που μπορεί να οδηγήσει αυτή η αιώνια απόπειρα εξαγοράς της ανάπτυξης. Δεν λειτουργεί πιθανότατα χρειάζεται ένα μοντέλο ανακατανομής στο μέλλον που θα λαμβάνει υπόψη αυτό το στοιχείο που ανέφερα. Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με το συμμετέχει κάποιο στο ευρώ ή όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει αυτό να αποφευθεί πάση θυσία. Αλλά λογικώ θα πρέπει να αποφευθεί να έχουμε μια Ευρώπη με πάνω από ένα νόμισμα. Είναι εκείνοι που δεν μπορούν να μπουν στο ευρώ ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ θα πρέπει αυτοί να επανεξετάσουν μακροπρόθεσμα τη θέση τους. Έρευνα και ανάπτυξη μετά. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος συντονισμός όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από ό,τι τώρα και θα πρέπει να συζητηθεί επίσης και μία μείωση συμμετοχής των κρατών μελών και αύξηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Ο κ. Κονφεράτη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι τα μεγάλα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν θα έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες επί του μέλλοντος της Ευρώπης. Αναφέρομαι λοιπόν στην κρίση στη Μεσόγειο που θέτει εκ νέου το θέμα της προμήθειας πρώτων υλών υπό διαφορετικές συνθήκες από ό,τι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια και αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία που θα οδηγήσει να εξετάσουμε πάλι σκοπιά την ενέργεια. Θα πρέπει να μειώσουμε το συναισθηματισμό αλλά και τα συναισθήματα μετρούν πολύ στη ζωή ενός ατόμου και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να συζητήσουμε τα θέματα της ασφάλειας και το πρόβλημα της ενεργειακής παραγωγής. Τώρα, στην παρούσα κατάσταση, επιβεβαιώνεται ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει ιδίους πόρους. Απλώς, με αυτόν τον απλό προϋπολογισμό δεν υπάρχει ελπίδα ανάκαμψης. Το θέμα των ευρωμολόγων και η φορολόγηση των χρηματοδοτικών συναλλαγών αντικειμενικά αποτελούν προτεραιότητα και για την Ένωση και για τα διάφορα κράτη-μέλη και μετά θα πρέπει να εντοπίσουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες των επενδύσεων. Και αν εντοπίσουμε τους πόρους θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι τα θεμέλια για την χρήση αυτών των πόρων. Πιστεύω ότι οι προτεραιότητες είναι δύο. Η πρώτη είναι η συμπλήρωση ενός δικτύου ε, υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλές ανισορροπίες μεταξύ διαφορών περιοχών της Ευρώπης και αυτό είναι βάρος της. Και όσον αφορά την ποιότητα της ζωής και όσον αφορά την έλκυση επενδύσεων διαφοροποίηση είναι καλή. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη γνώση. Το να γνωρίζει κανεί, η δασκαλία. Σε στιγμέ κρίση χρειάζονται επενδύσει στη γνώση και όμω η Ευρώπη κάνει ακριβώ το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι επένδυση στο σχολείο, ανεξάρτητα από τη μορφή του σχολείου, θα πρέπει να θεωρηθεί το σημείο αφετηρίας για να έχουμε ένα μοντέλο ανταγωνιστικό που ανταποκρίνεται στο όνομα, στον τίτλο αυτό. Ανταγωνιστικό μοντέλο. Ε, λοιπόν, τώρα καλώ τον συνάδελφο Βάιγκελ για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μύρο, η οποία όμως είναι πολύ επίκαιρη. Περί τίνος πρόκειται διότι κατόπιν των προσφάτων εξελίξεων που είχαν καταστροφικές διαστάσεις και λόγω αυτών των εξελίσεων η Ευρώπη έχει αναλάβει νέους νέα οικονομικά βάρη και όλοι ε, ζητούν να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη αλληλεγγύη και ειλικρίνεια. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για την αποκατάσταση του μηχανισμού και ε, των πηγών των ε, οικονομικών πόρων κατά τρόπον ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να συνδράμει και να επηρεάσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Η ερώτησή μου αναφέρεται σε μία ιδέα ενός νέου προγράμματος Marshall για τη Μέση Ανατολή διότι δεν βλέπω άλλη διέξοδο. Πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι μόνο χρηματοοικονομικό αλλά το οποίο θα περιλαμβάνει συγχρόνως και άλλες προσεγγίσεις, δηλαδή την κατάρτιση θεσμών και ε, ουσιαστικά κρατικού μηχανισμού. Θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για ένα δυνητικό πρόγραμμα Marshall, άλλοι το ονόμασαν πρόγραμμα Άστον ή και με διαφορετικές ονομασίες, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν πρέπει να είναι υπερβολικά φιλόδοξο και δεν θα πρέπει να εμπλέξουμε ή να εμπλακούμε στη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό αυτών οι οποίοι τις τελευταίες δέκα έχουν εποφεληθεί από τους ε, ιδιωτικούς ε, πόρους και αναφέρουμε εδώ στις πετρελοπαραγωγικές χώρες, ο κύριος Τσίλερ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους διάφορους εθνικούς βουλευτές που παρενέβησαν σήμερα και ο κύριος Μύροφ, ο οποίος έφυγε ίσως, αλλά νομίζω ότι τόνισε ότι η ενιαία αγορά, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες, δεν είναι ολοκληρωμένη μαζί και το ευρώ είναι πολύ μεγάλο για να αποτύχει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δύο είδη χωρών και ε, νομίζω ότι όταν ε, θα αντεπεξέλθουμε τις κρίσεις θα υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές από ό,τι υπήρχαν το 2004 διότι δεν θα υπάρχει μόνο η διαχωριστική γραμμή αυτών που είναι στην Ευρωζώνη και των άλλων αλλά ορισμένες χώρες θα ε, θα βρίσκονται σε ε, ένα χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο και στην Ευρωζώνη και εκτός διότι η διακίνηση των κεφαλαίων είναι συνδεδεμένη ε, και με το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος και όλα αυτά διασυνδέονται με τις διακρατικές χρηματοδοτήσεις. Οπότε ε, όσο και να αποπληρώνουμε τόσο περισσότερο θα πλουταίνουν αυτοί οι ε, οποίοι μας δάνεισαν και στις χώρες που πληρώνουν, ε, αποπληρώνουν θα χειροτερεύουν τα κοινωνικά προγράμματα και δεν θα υποφελούνται και αυτοί που ε, επενέδυσαν στις χώρες μας. Δεν θέλω εδώ να οξύνω τα πράγματα πολιτικά, νομίζω όμως ότι είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην καταστραφεί η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Χουντής για την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο πολύ να τους ευχαριστήσω για τις απόψεις και τα ερωτήματα που έθεσα. Αυτό αποδεικνύει κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι ότι υπάρχει εκτός των άλλων και μια κρίση νομιμοποίηση των πολιτικών που εφαρμόζονται. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος που παίζουμε εσείς σαν εθνικοί βουλευτές και εμείς σαν ευρωβουλευτές. Πάντως είμαστε εκ των υστέρων και σχολιάζουμε τώρα αν ήταν θετική ή αρνητική η απόφαση που ελήφθη προχθές για το λεγόμενο σύμφωνο για το ευρώ χωρίς να έχει προκύψει από πού νομιμοποιούνται οι κυβερνήσεις, χωρίς να διαβουλευτούν με τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και δεσμεύουν τις χώρες και τις οικονομίες τους με τόσο σκληρά μέτρα. Ο κύριος Μυρό λείπει κατά την ανάλυση του είπε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά έχουμε ορισμένους φραγμούς ακόμα. Και ακόμα σε κάποιο σημείο λέει επενδύουμε στην ευθεία του ιδιωτικού τομέα. Αν λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, το σύμφωνο για το ευρώ, αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο συνεχούς λιτότητας και περικοπής μισθών και δικαιωμάτων των εργαζόμενων, ας μην ψάχνει ο κύριος Μυρό πώ θα προκύψει η ανταγωνιστικότητα, α μην ψάχνει για διαφυΐα του ιδιωτικού τομέα. Αν συμπιέσει το εργασιακό κόστο, δεν θα πονοκεφαλιάσει πολύ να βάλει και καινούριε τεχνολογίε και καινούρια καινοτομία, τη αρκεί ότι θα έχει μεγαλύτερη ίσπραξη και μεγαλύτερη δυνατότητα κέρδου από τη συμπίεση του εργασιακού κόστου και την περιστολή των δικαιωμάτων, διότι αυτό είναι το μνημόνιο. Δεύτερο, σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα. Πού έχουμε φτάσει σήμερα, όπω σωστά είπε μια συνάδελφο πριν, η κρίση εμφανίστηκε ως κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, στη συνέχεια της πραγματικής οικονομίας, άρα και γιατί τα ξεχωρίζουμε. Και τέλος εμφανίζεται σήμερα ως κρίση χρέους, που όμως σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η κρίση του δημοσίου χρέους έχει αναγορευτεί στην αιτία τη κρίσης. Ότι αυτή φταίει για την κρίση. Και το ερώτημα που θέτω και όταν βρισκόμαστε μπροστά σε πρόεδρο τραπεζών. Πόση από αυτή τη ρευστότητα, τις ενέσεις που δόθηκαν στι τράπεζε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει πάει στην πραγματική οικονομία. Και δεύτερο, εφόσον στόχο μα είναι η απασχόληση, γιατί έχουμε την ανεργία να αυξάνεται στην Ευρώπη και έχουμε φτάσει στα 22 εκατομμύρια. Επομένω, μπορεί όλε αυτέ οι προθέσει, καλοπροαίρετε ακούγονται, μοιάζουν σαν, σαν την περίφημη στρατηγική τη Λισαβόνα που έλεγε για μια Ευρώπη ανταγωνιστική οικονομία και υπέσχετο πλήρη απασχόληση και είδαμε τα αποτελέσματα. Επομένως, νομίζω ότι λάθος βαδίζουμε. Η δική μας άποψη δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα που έχουν βγει για την κρίση, αλλά το θέμα είναι ότι και αυτές οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν θα μας φέρουν ούτε απασχόληση, ούτε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ρωτώ τώρα την Περβόνσου σαν εισηγήτρια αν θέλει να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το σύνολο των ε, συναδέλφων μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη συνδρομή του στην εργασία που έχουμε ξεκινήσει σε αυτή την ειδική επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε πλήρη διάταξη και από την αρχή της θητείας μας ε, είχαμε πολλές ανταλλαγές. Ήρθατε εδώ, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε, απαντήσατε στα ερωτήματά μας μας στηρίξατε την ε, ε, ε, έκθεση την οποία υιοθέτησε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο πέρυσι και όπως είπε ο κύριος Μύροφ δεν πρόκειται να υπάρχει διέξοδος από την κρίση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν εσείς και εμείς από κοινού μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναβιώσουμε την πίστη ε, στο ότι απέναντι στην παγκοσμιοποίηση χρειαζόμαστε μία ενωμένη Ευρώπη. Τη στιγμή όμως όπου ο νότος της Μεσογείου μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι οι αξίες μας, η προσμονή ελευθερίας και κράτους δικαίου πρέπει σαν κοινοβουλευτική να εφαρμόζουμε τις αρχές αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές πιστεύουμε ότι υπάρχει μία παρεκτροπή με υπερβολική κυβερνητική παρέμβαση η οποία επιβάλλεται και αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον μας αυτών των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και των πολιτών της Ενώσεως. Ο πρόεδρος Μίροφ ε, είχε επέμβει στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στην έκθεση την οποία υιοθετήσαμε μετρήσαμε πόσο η έξοδος από την κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν στη δυνατότητα ανακάμψεως και χρηματοδοτήσεως με ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις μακροπρόθεσμες. Και επ' αυτού θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις κατόπιν των σχολείων που προηγήθηκαν. Ο πρόεδρος Μύροφ είπε ότι χρειαζόταν μία νομική ασφάλεια και το κατανοούμε. Αλλά εγώ εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι πολλές φορές πρόκειται για επενδύσεις πολύ καπιταλιστικές τις οποίες εάν δεν προσέξουμε δεν θα μας επιτρέψουν μόνο να λύσουμε τα προβλήματα απασχόλησης που αντιμετωπίζουμε. Άρα οι ε, διατυπώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας όπως το επαναλάβαμε πέρυσι τον Οκτώβριο με το άρθρο 9 μας ζητούν να εξετάσουμε όλες τις δημόσιες πολιτικές των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις. Όχι μόνο για να κάνουμε ε, μία μελέτη των επιπτώσεων όπως κάνουν ορισμένα γραφεία αλλά για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δημιουργία θέσεων εργασίας. Ορισμένοι είπαν ότι ανησυχούν πάρα πολύ για τις ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες συζητούνται για τις χρηματαγορές και η εντύπωση την οποία αποεκόμισα από πολλά σχόλια ήταν ότι από τη μια πλευρά θα υπήρχε μεταρρύθμιση των χρηματαγορών και δεύτερον από την άλλη πλευρά της ανάγκης ε, ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και ε, την ε, ενόχληση ότι δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο θέματα. Συμφωνώ με την ανησυχία και συνολικά εγώ ανησυχώ γιατί πολλές φορές νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει ε, μία μεταρρύθμιση βάση καταλόγου και όχι προγράμματος. Αυτό θίξαμε και στην έκθεση που καταρτήσαμε διότι πολλές φορές αφήνουμε τους ε, παίκτες της αγοράς να ε, διαμορφώσουν την αγορά σύμφωνα με τις ανάγκες τους αντί να αναπροσανατολίσουμε ε, τις χρηματαγορές της Ευρώπης βάσει των πραγματικών αναγκών. Και ε, θα έπρεπε μια τέτοια συζήτηση να γίνει ίσως στο G20 αλλά και εις ε, την Ευρώπη διαπιστώνω ότι δεν γίνεται επαρκώς η εξέταση αυτή. Και η Βασιλεία 3, ή άλλες συμφωνίες για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των αναγκών δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς. Μακροοικονομικά πολλοί αναφέρθηκαν στις ανισότητες που υπάρχουν παγκοσμίως και εγώ θα ήθελα να παρέμβω σε ένα θέμα που μου φαίνεται πολύ ουσιαστικό. Ότι δηλαδή μετά από την κατάρρευση της Lehman Brothers ορισμένοι είπαν ότι έπρεπε να προσθέσουμε στο θέμα της σταθερότητας των τιμών τη σταθερότητα των χρηματαγορών. Αλλά πέραν τη σταθερότητα των χρηματαγορών, πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα διεξάγεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ε, αν ε, συμβάλλει εις ε, μακροοικονομικές αστάθειες, διότι έρχομαι από μία χώρα όπου οι εξωτερικές άμεσες επενδύσεις πάντοτε μετρώντουσαν σαν αποτέλεσμα το θελκτικότητος της οικονομίας της χώρας μου αλλά αυτό προκαλεί κερδοσκοπία και ε, υπάρχουν και επιρροές ε, εις ε, την αγορά παραγωγής που πάντοτε δεν είναι προς τον των τοπικών ενδιαφερομένων. Υπάρχουν υπερβολικές αποδόσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τους στόχους τους οποίους επιζητούμε όταν εμείς σκεφτόμαστε τις ανάγκες της πραγματικότητας οικονομίας. Δύο τελευταίες παρεμβάσεις. Ορισμένοι έκαναν μία έκκληση για την εσωτερική αγορά. Ε, είπαν και όντως συμφωνώ ότι είναι ένα κοινό αγαθό της Ευρώπης και ε, μεταξύ την ανάκαμψη δια της εσωτερικής αγοράς και της ευρωπαϊκής αγοράς ενεργείας προτιμώ τη δεύτερη παρόλο που πρέπει να σέβεται και την εσωτερική αγορά. Τουλάχιστον στο θέμα της ενεργείας π.χ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Έγγελς όταν είπε ότι το θέμα της έμονης ιδέας της αναπτύξεως δεν πρέπει να τοποθετείται όπως είναι και παρόλο που είναι εκπρόσωπος του ΕΛΚ ελπίζω ότι στο τέλος θα συμφωνήσουμε και σε αυτό το σημείο όταν λέει ότι πέραν της αναπτυξής θα πρέπει να κοιτάξουμε την κατανομή γιατί υπάρχει μια διαφορετική πρόκληση και πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα της φορολογίας. Πολλοί το ανέφεραν και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα αυτού του Σαββατοκύριακου ακόμη θα πρέπει να υλοποιηθεί. Αλλά ευχαριστώ για την πρώτη ανταλλαγή που είχαμε και που θα ενσωματώσουμε μέχρι τον Ιούλιο στην τελική μας έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της ε, σημερινής μας ε, συνεδριάσεως η οποία έχει σαν κύκλο επενδύοντας στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του 2020 και ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Φίλιπ Μάισταρ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το Λουξεμβούργο ο οποίος τώρα ανεβαίνει στο Προεδρείο και είναι ε, πρόεδρος ε, ήδη από το 2006 οπότε επεκτάθη, ε, το, παρετάθη το, η εντολή του για άλλα 6 χρόνια και προηγουμένως ήταν επί 10 χρόνια Υπουργός Οικονομικών στο Βέλγιο το 1990 ήταν, είχε ανακηρυχθεί από το περιοδικό Euro Money ο Υπουργός Οικονομικών της χρονιάς. Ε, και ολοκλήρωσε την καριέρα του την πολιτική σαν αντιπρόεδρος του κρατηδίου της ε, ε, χώρας του. Χαίρομαι λοιπόν που θα προεδρεύσει, θα, θα κάνει την εισαγωγή και την κεντρική ομιλία για τη δεύτερη συνεδρίαση και του δίνω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου καταρχά να σας πω πόσο με τιμά αυτή η ευκαιρία που έχω στη διάθεσή μου να μιλήσω στην Επιτροπή σας, η οποία συζητεί κρίσιμα προγράμματα για το συλλογικό μας μέλλον και έχει μια σύνθεση που προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι συναθρίζει και Ευρωπαίους βουλευτές, αλλά και εθνικούς, τουλάχιστον για τη σημερινή συνεδρίαση. Δεν θα επεκταθώ επί μακρόν Επί του τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ξέρετε ότι είναι η Τράπεζα των Κατώμερων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θεσπίστηκε από τι συνθήκε σαν αποστολή δυνάμει των συνθήκων την υποστήριξη την οικονομική των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εκείνου που θέλουν να γνωρίζουν περισσότερο όσο αφορά το ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόσφατα, μπορούμε να διανύμουμε ένα σημείωμα που περιγράφει τη συνεισφορά μας στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη που εθέτηκε το Δεκέμβριο του 2008. Βλέπετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνέβαλε στην προσπάθεια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ όμω σήμερα ε, επί των θεμάτων που θίξατε. Ποιο είναι ο ρόλος δηλαδή των επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη του 2020. Θα ήθελα να ξεκινήσω μέσω σύντομης υπενθυμίσεως της σημασίας των επενδύσεων για την ανάπτυξη. Εν γέννη αναγνωρίζεται ότι η διαμόρφωση σταθερού κεφαλαίου και η διαμόρφωση του αποθεματικού από μαζί δημιουργούν την επένδυση όπως αναφέρεται παραδοσιακά και είναι σημαντικός παράγων για τη συγκυριακή ανάπτυξη και τις συγκυριακές εξελίξεις. Και έχει σημαντική συνέπεια η επένδυση επί της διαμόρφωσης του ΑΕΠ. Αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι είναι σημαντικό και πέρα από τους κύκλους τους οικονομικούς, διότι η επένδυση ε, είναι κρίσιμη για την καινοτομία και την παραγωγικότητα και για το δυναμικό, το αναπτυξιακό της οικονομίας. Έχετε εδώ ένα γράφημα που σας δείχνει ότι πράγματι στην κρίση που περνάμε η δραστική πτώση των επενδύσεων έχει μεγάλη σημασία και συμβάλλει τα μάλα για τη μείωση του ΑΕΠ. Βλέπετε στο γράφημα το γκρίζο είναι η διαμόρφωση του σταθερού κεφαλαίου που μειώνεται και η διαμόρφωση του αποθεματικού, η διαφορά του αποθεματικού. Και η ύφεση του 2009 εξηγείται κατά πολύ από τη μείωση των επενδύσεων. Το 2010 η διαμόρφωση σταθερού κεφαλαίου συνέβαλε κάπως, άλλαξε κάπως με αρνητικό πρόσημο, θα είναι θετική εξέλιξη όμως φέτος. Αυτό καταδεικνύει πως οι επενδύσεις σημαντικές. Και ακόμα και αν μπορούμε να περιμένουμε μια ανάκαμψη φέτος, όμως παρόλα αυτά το αναπτυξιακό δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας που ήδη ήταν πάρα πολύ χαμηλό πριν από την κρίση, επηρεάστηκε αρνητικός από αυτή την πτώση τη μεγάλη των επενδύσεων. Συνεπώς, το ερώτημα που θέσατε κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκόπιμο και σχετικό πώς μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις που είναι αναγκαίες ούτως ώστε να αυξηθεί το δυναμικό αναπτύξεως των ευρωπαϊκών οικονομιών κάτι που στο κάτω-κάτω αποτελεί τον σημαντικότερο στόχο της στρατηγικής Ευρώπη για το 2020. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τη μια επενδυτικές ανάγκες τεράστιες. Τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις και στα νέα κράτη-μέλη και στα πιο παλιά. Και για τη δημιουργία νέων υποδομών, αλλά και για τον εξυγχρονισμό των υφισταμένων υποδομών, εκτιμήσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε, ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη του 2020 θα χρειαζόταν μια επένδυση σε υποδομές ανάμεσα στο 1,53 και 2,3 ευρώ από τώρα μέχρι το 2020. Άρα πάνω από 2 ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ και να προσθέσουμε και τις επενδύσεις σε άλλους τομείς πέραν των υποδομών και κατά την άποψή μου εξίσου σημαντικούς. Άρα τεράστιες ανάγκες υπάρχουν για επενδύσεις. Βλέπουμε ποιες είναι οι πηγές χρηματοδοτήσεως. Οι πηγές τείνουν να στερεύουν. Γιατί? Διότι άφησε τα ίχνη της η κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα Υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί φορείς που εξαφανίστηκαν, όπως η ασφαλιστική μόνο online, online μάλλον. Οι τράπεζες προχωρούν όλο και πιο προσεκτικά σήμερα και οι νέοι κανόνες της Βασιλείας τρία δεν ενθαρρύνουν σίγουρα τις τράπεζες να διανοδοτούν περισσότερο και από μακροπρόθεσμα και να αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους. Άρα τι αναμένουμε. Περιμένουμε η τραπεζική χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα παραμείνει σχετικά περιορισμένη για τα επόμενα χρόνια. Και μετά γνωρίζετε ποιοι είναι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Υπάρχουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν σημαντική αύξηση των κονδυλίων των προπολογισμών τα επόμενα χρόνια. Άρα έχουμε τεράστιε ανάγκε χρηματοδοτήσει από τη μια, ένα τραπεζικό τομέα που ακόμα είναι εύθραυστο και αντιμετωπίζει νέου κανόνε συνετή διαχειρίσεω και θα έχει την τάση να μειώσει τι μακροπρόθεσμε υποχρεώσει και δεσμεύσει πιο επικίνδυνε, δημοσιονομικού περιορισμού μεγάλου. Πώ να συμφιλειωθούν αυτά τα διάφορα στοιχεία. Παρά μόνο προσπαθώντας να βρούνε κάποια, κάποιο καταλήτη και αποτελέσματα μόχλευσης συνδυάζοντας το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα χρηματοδότησης. Και σε αυτή την παρουσίαση ήθελα να επιμείνω ενδεχομένως επί του, φαινομένου μοχλεύσεως που μπορεί να, να πορεύσει από την κοινή δράση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η χρήση επιδοτήσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν επαρκές κέρδος, ε, ανεπαρκές κέρδος είναι σπατάλη χρημάτων. Αντιστρόφως, η χρήση να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δάνεια τραπεζικά για επενδύσεις που είναι πολύ χρήσιμες για την οικονομία μεν, αλλά έχουν απόδοση εσωτερική οικονομική πολύ χαμηλή, είναι και αυτό μια αυτοπάτη. Συνεπώς, θεωρούμε ότι μεταξύ εκείνων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, χρηματοδοτηθούν μέσω των εμπορικών τραπεζών, λόγω περιορισμένου κινδύνου, λόγω επαρκούς αποδόσεως και στο άλλο άκρο αυτό που έχει χρηματοδοτηθεί από επιδοτήσεις, διότι προφανώς ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος ή η απόδοση είναι αρνητική. Υπάρχει ανάμεσα στα δύο μια διάμεση περιοχή, ζώνη, όπου εκεί η κοινή δράση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υλοποιήσουν κάποια προγράμματα, όπως λέμε στην ορολογία μας. Δηλαδή, να, είμαστε, ε, να έχουμε τη δυνατότητα, είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες και από τα δάνεια. Είναι αυτή, ε, σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη που θέλω να επικεντρωθώ σε αυτή τη φάση της παρέμβασής μου. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς κάτι, να σας αναφέρω τι ήδη έχει πραγματοποιηθεί, ποια είναι τα κοινά, τα μεικτά μέσα που έχουμε υλοποιήσει με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφερόμενος επίσης και σε κάποιες μελλοντικέ προσεγγίσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμορφώσαμε δύο κοινά μέσα η εργαλεία. Το πρώτο είναι το, το μέσο για την έρευνα, για το, για το μερισμό του κινδύνου και το άλλο ένα σύστημα εγγυήσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Καταρχάς, το πρώτο το μέσο για την έρευνα που ανέφερα είναι κοινή η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συναθρίζοντας εκεί, σε αυτό το μέσο, ένα ποσό από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ένα ποσό που πήραμε από το ετήσιο κονδύλιο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργούμε ένα απόθεμα, αν θέλετε, ένα ποσό που επιτρέπει, μια πρόβλεψη, αν θέλετε, για να χρηματοδοτεί η τράπεζά μα ερευνητικά προγράμματα ε, πιο επικίνδυνα και προγράμματα αναπτυξιακά. Αυτό ξεκινήσαμε εδώ και μερικά χρόνια να το κάνουμε και έγινε μια αξιολόγηση από ομάδα ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων και αυτή η αποτίμηση, η αξιολόγηση παρουσιάστηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν θετικά τα απορίσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται αυτή τη θετική άποψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου που μας πέρασε συνέστησε αυτή η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και την περασμένη εβδομάδα ψήφισε ένα ψήφισμα προς την ίδια κατεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε ένα κοινό μέσο λοιπόν που θα επιτρέψει να έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο, το φαινόμενο μόχλευσης. Το τέλο του περασμένου έτου, είχαμε δώσει κάποια δάνεια, εγκρίναμε κάποια δάνεια για 6,3 δις ευρώ που χρηματοδότησαν επενδύσει τη τάξη των 16 δι, άρα ήδη έχουμε το φαινόμενο μόχλευση και όλα αυτά χάρη σε μια παρέμβαση του ευρωπαϊκού προπολογισμού τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπετε το παραπιστικό φαινόμενο. Από 300 εκατομμύρια ευρώ του ευρωπαϊκού προπολογισμού μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε επενδύσει για ένα συνολικό ποσό 16 δισεκατομμύριων. Γιατί? Διότι αυτή η επένδυση, αυτή η παρέμβαση του ευρωπαϊκού προπολογισμού επιτρέπει να επιμεριστεί ο κίνδυνο να τον μοιραστούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άρα μειώνεται η κατανάλωση κεφαλαίου για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα ενό υπάρχοντος μέσου και το οποίο δίνει αποτελέσματα. Το δεύτερο εργαλείο, το δεύτερο μέσο είναι πιο καινούριο, πιο πρόσφατο. Είναι το σύστημα των εγγυήσεων για ένα συγκεκριμένο είδος κινδύνου που γνωρίζουμε με, τα νέα, με τις νέες υποδομές των μεταφορών. Δηλαδή, όταν το εισόδημα που δημιουργείται από την υποδομή τα πρώτα χρόνια της εκμετάλλευσης δεν είναι στο επαρκέ στο αναμενόμενο επίπεδο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα. Είναι ένα σύστημα λίγο πιο περίπλοκο, αλλά στο τέλο επιτρέπει σε εμπορικέ τράπεζε να συνεχίζουν να δανοδιοτούν εκείνους που προωθούν προγράμματα έργα υποδομών με την εγγύηση ότι αν κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών εκμεταλλεύσεως τα εισοδήματα δεν είναι επαρκή, και δημιουργούνται δυσκολίε για εκείνου που υλοποιούν το έργο και δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό του, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντικαθιστά την Εμπορική Τράπεζα, γίνεται υποκείμενο δανειοδότη εκείνου που εφαρμόζει το υλοποιεί το έργο, με τη δυνατότητα καλύψή περιορισμένη στην αρχή του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Άλλο ένα, μεικτό, άλλο ένα παράδειγμα μεικτού εργαλείου. Εάν έχουμε, εξετάσουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές στρατηγική του 2020, δεν θα πρέπει να επανεφεύρουμε απαραίτητα τον τροχό. Επί τη βάση των πρώτων παραδειγμάτων μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα, να πάρουμε μαθήματα και έχουμε κοινό συμφέρον να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κοινά εργαλεία, κοινά μέσα, σχετικά απλά στην εφαρμογή τους, αυτό είναι σημαντικό, τα οποία μέσα θα έχουν εξελισσόμενο χαρακτήρα, θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται άμα θέλετε. Αυτό που επιστρέφει θα μπορούμε να καλύψουμε διάφορους τομείς και αυτά τα μέσα θα οδηγήσουν μεγαλύτερη ορατότητα των έργων, των δράσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί το χαρακτηριστικό των νέων χρηματοπιστωτικών αυτών εργαλείων, των μέσων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν παρουσίασα. Ένα από τα νέα μέσα, τα νέα εργαλεία τα οποία εξετάζουμε είναι τα, τα project bonds, τα διάφορα αξιόγραφα, τα ομόλογα που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα έργα. Μπορώ να απαντήσω εγώ τις ερωτήσεις. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν. Ξεκινήσαμε από μια διαπίστωση που ήδη ανέφερα. Τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις, τις μεταφορές, την ενέργεια, ε, της ευρυζωνικής. Ξέρετε τα στοιχεία για να πετύχουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών, να τα υλοποιήσουμε. Και θυμάμαι ότι ο πρόεδρος Ντελόρ ξεκίνησε αυτή την ιδέα των διευρωπαϊκών δικτύων, την έριξε αυτή την ιδέα, για να ολοκληρώσουμε τα δίκτυα χρειαζόμαστε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Ταυτόχρονα λοιπόν, όπως ανέφερα, δημόσιοι προπολογισμοί είναι περιορισμένοι, οι τράπεζες είναι πιο διστακτικές να υπομιστούν μακροχρόνιους κινδύνους και ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείε monoline που εξαφανίστηκαν ή μειώθηκε πολύ η μειωθηκε πολυ θεση τους. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Διότι αυτές οι ασφάλειες monoline έδιναν στα ομόλογα που εξέδιδαν οι, ε, οι εταιρείε που εξελούσαν έργα έδιναν ε, τη δυνατότητα, την εξασφάλιση να έχουν να αποκτήσουν αξία και να αξιόπιστα αυτά τα ομολόγα. Άρα θέλουμε να ελκύσουμε, προσελκύσουμε ιδιωτικού πόρου επιτρέποντα εταιρείε που υλοποιούν έργα να εκδίδουν ομόλογα τα οποία θα έχουν τέτοια ποιότητα τα ομόλογα που θα μπορούν να αγοραστούν από τους θεσμικούς επενδυτές, συνταξιωτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και όλα αυτά εδράζονται επί της ιδέας του trenching, δηλαδή να δημιουργούνται trenching μάλλον ε, στιβάδες στο χρέος θα υπάρχει το senior, το πάνω, το, το κυρίως ε, χρέος που θα έχει τα επαρκή εχέγγια για τους επενδυτές για να μπορούν να αγοράζουν τα ομόλογα. Άρα έχουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τάπεζας Επενδύσεων, η οποία γίνεται αυτή η παρέμβαση στο επίπεδο που βλέπετε στο γράφημα, στο μεσαία, στη μεσαία στιβάδα, υπό τη μορφή ε, υποκειμένων ε, αξιογράφων και Τέλο που θα πούμε σε λεπτομέρειε. Η Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων δίνει ένα δάνειο υποκείμενο που ακριβώ επειδή είναι υποκείμενο δίνει ένα χαρακτήρα υψηλότερο senior στο τμήμα του χρέους που αποτελεί αντικείμενο της έκδοσης των ομολόγων για το συγκεκριμένο έργο. Άρα ένας μηχανισμός αυξήσεως της πίστοσης, ανα, αναβάθμισης της πίστοσης η επένδυση του ευρωπαϊκού προπολογισμού επιτρέπει τον επιμερισμό του κινδύνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο πολύ περιορισμένο από την αρχή. Δεν θα έρχει contingent liability για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ευθύ εξ αρχή θα ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγιστο δυνατό κόστος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και αν παρελπίδα το κόστος μεγαλύτερο, αυτό, η διαφορά του κόστους θα αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πάνω σε αυτό το σχέδιο κινούμεθα και εργαζόμαστε. Ξεκινήσαμε με δημόσια διαβούλευση και περιμένουμε να αντιδράσεις. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε το ιδιωτικό τομέα είναι θετικότατες. Άρα είναι ένα μέσο αυτό για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε και άλλη ιδιωτική χρηματοδότηση για έργα υποδομών. Αναφέρθηκα στο επίκαιρο αυτό παράδειγμα, επειδή είναι επίκαιρο, αλλά υπάρχουν ε, σαφώς και άλλα εργαλεία και άλλα μέσα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντά σα τι πιστεύω, ότι η επόμενη δεκαετία πιστεύω θα είναι κρισίμου σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώ η Στατηγική Ευρώπη του 2020 θεωρώ ότι είναι ουσιοδέστατη, είναι πάρα πολύ σημαντική εάν θέλουμε να αυξήσουμε το δυναμικό, το αναπτυξιακό της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι ξεκάθαρο ότι απαιτούνται επενδύσεις και όχι μόνο στις υποδομές όπως ανέφερα, αλλά χρειάζονται και επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των πτυχιούχων της ανωτέρας εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα, είναι κεφαλαιούδου σημασία. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην καινοτομία, θα πρέπει πολύ πιο γρήγορα να διαδίδεται καινοτομία σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι σημαντικό άξονα τη στρατηγική Ευρώπη του 2020, αλλά είναι σαφέ επίση ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσει και τα εθνικά κοινοβούλια να φροντίσουν αυτή η στρατηγική να γίνει δική του, να την εστερνιστούν, να τη δεχτούν. Να δεχτούν επίση έναν καλύτερο συντονισμό σε μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση η οποία θα είναι ενισχυμένη. Θεωρώ ότι είναι προαπαιτούμενο αυτό για την επιτυχία της στρατηγικής. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι συζητήσεις στην Επιτροπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν άμεσα και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Διότι δεν θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε σωστά την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 αν οι κυβερνήσει και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν εμπλακούν πλήρω αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Μάιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας για την εξέβρεση συνένεσης με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο ότι και εμείς είμαστε απόλυτα απεπισμένοι ότι αν δεν υπάρχει απόλυτο συντονισμό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε τους φιλόδοξους αυτούς του στόχους. Θα ακολουθήσουμε όπως και την πρώτη φορά την εξή διαδικασία. Θα καλέσω καταρχάς τους εκπροσώπους των χωρών ε, ε, της Τρόικας. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον κύριο Έκερς. Έχετε τρία λεπτά maximum. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συμφωνήσω με αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος, ότι δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, με τα εθνικά κοινοβούλια. Χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα των ε, της πατάλης και το θέμα των αποδόσεων των επενδύσεων των τελευταίων χρόνων. Η καινοτομία, η έρευνα και η εκπαίδευση αποτελούν τους πιο σημαντικούς τομείς. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο θα καταστούμε ανταγωνιστικοί στους, σημαντικούς, στους τομείς αυτούς. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι η ενέργεια, οι πόροι και οι πρώτες θα πρέπει να σκεφτούμε όχι κοντόφθαλμα, αλλά μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλογιστούν σε ποιου τομεί. Όσο εθνικά κοινοβούλια μπορούν να πετύχουν τους ε, πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους και σε ποιους τομείς θα πρέπει να διατυπώσουν ευρωπαϊκούς στόχους. Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά και την φορολογική πολιτική. Κοιτώντας τι γίνεται και πού πραγματοποιούνται οι πιο πολλές επενδύσεις στην Ασία, είναι μάλλον στην Ασία και στην Κίνα, αυτά που ακούσαμε εδώ είναι βασικά το κατά πόσον υπάρχει κάποια ανάλυση σχετικά με την εξάρτηση της Ευρώπης από τους τομείς αυτούς, κατά πόσον υπάρχει όφελος για την Ευρώπη και κατά πόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε την ανάπτυξη αυτή και πού μπορούμε να σημειώσουμε καλύτερες επιδόσεις. Θεωρώ ότι η στρατηγική για το 2020 είναι πάρα πολύ σημαντική υπό την έννοια ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια συνένεση στο εσωτερικό της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τα θέματα περιφερειακών επενδύσεων, θέματα σπατάλης και σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα και αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να καταστεί πιο αποδοτική και πιο ανταγωνιστική. Αυτά λοιπόν ήθελα εν συντομία να αναφέρω στο δεύτερο τμήμα της ε, συνεδρίασης. Θα ήθελα να πω επίσης ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ανέφερε ο Πρόεδρος ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος χρόνου και ότι πραγματικά χρειαζόμαστε πιο πολύ συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια για την επίλυση των ζητημάτων του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα επόμενος ομιλητής. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μέιστατ για την παρουσίασή σας. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η χώρα μας έχει υποστηρίξει πλήρως και υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της Ευρώπης της 2020 και δεδομένη και της ένταση που περιγράφεται ότι επικρατεί κύριε Μέιστα μεταξύ τη ανάγκη για επενδύσεις και κατά δεύτερον της, του ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών, να σας πω ότι αυτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Μία ε, παρατήρηση και μία ερώτηση. Αυτή η άσκηση ισορροπίας ε, μετακυλείται από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και αντιστρόφως. Βασίζεται ουσιαστικά στα εθνικά σύνορα και νομίζω θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η οικονομική πραγματικότητα δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα αλλά επικρατούν ουσιαστικά τα οικονομικά κλάστερ τα οποία δεν σέβονται τα εθνικά σύνορα. Έχουν δική τους αυτονομία και δυναμική. Θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε λοιπόν αυτά τα περιστατικά, αυτά τα γεγονότα σε περίπτωση που τεθεί κάποιος έλεγχος από πλευράς εθνικών κρατών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η Ευρώπη κατά την εξολόγηση των εθνικών εκθέσεων να ε, διευκρινίζει το περιφερειακό επίπεδο και επίσης τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάλυση σε εθνικό επίπεδο μπορούν να καταλήξουμε, μπορεί να οδηγήσουν αυτές οι αναλύσεις σε συστάσεις αντιπαραγωγικές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τη σημασία εκ νέου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συχνά αποτελούν ε, πηγές ε, σημαντικές για την οικονομικό ιστό της κοινωνίας, παρέχουν θέσεις εργασίες ασφαλής και επίσης ε, για τη μεταρρύθμιση της Βασιλείας 3 να μην αποβεί εις βάρος της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των βελγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι δεν φτάνει επαρκώς τις επιχειρήσεις που αποτελούν το στόχο της. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια εγγύηση του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί για περιφερειακό ταμείο και όχι μόνο για ομοσπονδιακό ταμείο συμμετοχή. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, ο κύριο Κλάινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Φίλιπ Μάιστατ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μας μιλάει και μας αναφέρει κάποιες καλές ιδέες σε εποχές κρίσεων, σε εποχές που θέλουμε να ξεπεράσουμε και να επικοινωνήσουμε την κρίση. Ζούμε σε εποχές λιτότητας, οπότε αναγκαστικά πρέπει να σκεφτούμε σε κάθε χώρα και σε κάθε επιχείρηση τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Όλες οι προτάσεις λοιπόν που μας υποδεικνύουν έναν τρόπο επίλυσης των προβλημάτων και το πώς μπορούμε να βρούμε νέες επενδυτικές λύσεις είναι σημαντικές για μας. Για την Πολωνία, η οποία διέρχεται τα τελευταία χρόνια επίσης μια σημαντική κρίση, αλλά και ως μοναδική χώρα στην Ευρώπη με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, πρέπει να πούμε ότι μας απασχολούν τα θέματα αποταμίευσης και της μείωσης ε, των έλλειμμάτων ε, προϋπολογισμού. Και γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις σας είναι τόσο ενδιαφέρουσες, γιατί καταδεικνύουν ότι παρά τα οικονομικά προβλήματα μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα μέσα επενδύσεων που έχουμε στην διάθεσή μας για μας τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην ε, απαρνηθούμε την αρχή της αλληλεγγύης και να μην της ελαχιστοποίησης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Τις επενδύσεις λοιπόν στην ενέργεια, την επένδυση, την εκπαίδευση συγγνώμη, και τις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά για εμάς για το πώς πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Οι ιδέες σας είναι πάρα πολύ ωφέλιμες και ασφαλώς και θα τις αξιοποιήσουμε και ασφαλώς θα σας πούμε και τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τις οποίες λάβαμε, η ομιλία του κ. Μάιστατ και η αναφορά στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες αλλά και στα παλαιά κρατημέλη. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, καταλαβαίνουμε ότι οι επενδύσεις και στα νέα αλλά και στα παλαιά κράτη-μέλη αποτελούν τον κινητήρα της μελλοντική οικονομίας, μιας οικονομίας η οποία θα μας ε, βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσης θα αποτελέσουν ένα είδος κινητήρα για την ανάπτυξή μας. Υποστηρίζουμε απόλυτα λοιπόν τις προτεραιότητες αυτές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική της Ευρώπης το 2020. Γι' αυτό λοιπόν οι ιδέες που συζητούμε εδώ μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι τόσο σημαντικές για εμάς και μας δίνουν και μια καλή προοπτική για μελλοντικέ λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσικάνε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δύο λεπτά. Thank you very much. Indeed. Ευχαριστώ. Όντως συζητάμε περισσότερο για τη σταθερότητα και θα έπρεπε να μιλάμε για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από το σύμφωνο σταθερότητος σωστή σύμφωνο βιωσιμότητος και αναπτύξεως ε, όπως ε, είπαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και της Τράπεζας Επενδύσεως, βασικό στοιχείο είναι τα κεφάλαια και τα κεφάλαια κινδύνου που θα πρέπει να συμβάλλουν στην σε καινοτόμες ε, τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στην κοινωνία. Ε, επίσης ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν φιλόδοξοι στόχοι ε, όχι μόνο στο περιβάλλον ε, και στην κοινωνία αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και ένα, μια εποπτεία για το περιβάλλον των επενδύσεων για να επιτύχουμε. Ένα άλλο θέμα είναι οι προπολογισμοί οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αμφιλεγόμενες δραστηριότητες θα πρέπει εφόσον έχουμε περιορισμένους πόρους να τους χρησιμοποιήσουμε για μεγαλύτερη ανάπτυξη, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να υπάρχει και μία λογιστική των διαθέσεως των πόρων αλλά χρειαζόμαστε συγχρόνως συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι σημαντικά και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μία διαφοροποίηση προς την ίδια κατεύθυνση. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξέρω εάν ε, μπορεί να σχολιάσει ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Επενδύσεων για τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε για τα κεφάλαια κινδύνου και είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα υπάρχουν τρεις ε, ομιλητές, ε, ο κύριος Χάρισον από τη Βουλή των Λόρδων, ο κύριος Ροζέτη Ιταλός και ο κύριος Κόλα από τη Σλοβακία. Καταρχήν όμως ο κύριος ε, Χάρισον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ε, μεγάλη χαρά που σας υποδεχθήκαμε στη Βουλή των Λόρδων που τώρα ε, θα δημοσιεύσει την έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και εκεί βασίζονται και τα σχόλιά μου διότι τονίζουμε την σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τον προϋπολογισμό να δούμε πού μπορούμε να επηρεάσουμε τις μεταφορές την υγεία εγώ θα επανερχόμουν στο προϋπολογισμό από μηδενικής κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ε, προσαρμόσουμε και τις πιο φτωχές χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε συγχρόνως μεγαλύτερη ευελιξία στον προπολογισμό μας κατά τρόπον ε, όταν ε, θα εξέλθουμε από ε, την περίοδο στενότητας που περνάμε τώρα να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη και θα πρέπει ακόμη να αναμένουμε την ενιαία αγορά και περιμένουμε ακόμη ακόμη να δούμε πώς η αγορά αυτή θα μπορέσει να είναι φιλική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις διότι θα πρέπει η στρατηγική για το 2020 να είναι βελτιωμένη σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας που δεν επέτυχε όπως ελέγχθη επανειλημμένος. Ένα άλλο θέμα είναι πώς ο, ο Επίτροπος Ντεγκούχτ ε, θα δημιουργήσει δημοσιεύσει σχόλια για το διεθνές εμπορόριο όπου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο επιθετική και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας και τέλος ε, όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα θέλω να σας πω ότι η μελέτη μας θα έχει ολοκληρωθεί τέλος Μαρτίου και με τα χαράς θα αποστείλω σε όλους σας αντίγραφα για να ε, συμπεριλάβετε στη στρατηγική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Ο κ. Τζοτζέτη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι υπάρχει δυσαναλογία μεγάλη μεταξύ των φιλόδοξων στόχων που θέτουμε με στρατηγική το 2020 και των απαντήσεων που κατορθώνουμε να δώσουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό σε αυτού του είδους την πρόκληση. Ο πρόεδρος Μαϊστάτ, κατά την άποψή μου, διευκρίνησε, ξεκαθάρισε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αναγκών και των πόρων. Όσον αφορά των δημοσίων πόρων, η δημοσιονομική πειθαρχία που έχουμε θεσπίσει δεν κάνει διάκριση μεταξύ τρεχόντων δαπανών και επενδύσεων. Δεν μπορούμε να βραβεύσουμε, αν θέλετε, την ποιότητα της δαπάνης. Και απ' την άλλη δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποια απάντηση πιστική και οριστική στη, τη μοναδική πραγματική απάντηση, ανά απόψή μου, στις, στα ευρωμόλογα που καλύπτουν τι ανάγκε στο δημόσιο τομέα. Όσον αφορά τους ιδιωτικούς πόρους, χρηματοδοτήσεω, νομίζω θα πρέπει να γίνει δελεχή προβληματισμό από αυτών που συμβαίνουν και προωθούνται μέσω τη Βασιλεία 3, διότι η Βασιλεία 3 αυξάνει το, την ανάγκη κεφαλοποίησης των, των τραπεζών, του αποθέματος και ίσως τελικά μέσω αυτών των πιο αυστηρών προδιαγραφών να βρεθούν σε δυσχερή θέση μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι θα είναι πάρα πολύ ε, προσεκτικές οι τράπεζες και μετά και επιχειρήσεις. Η Βασιλεία 3 θα έπρεπε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καταπολεμήσει και παρκώς και την κερδοσκοπία των τραπεζών όσον αφορά τα παράγωγα. Χρειάζεται προσοχή στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Επενδύσεων που είναι στη φαιά αυτή ζώνη που είπε πολύ σωστά ο μιλητής μεταξύ των επενδύσεων που χρηματοδοτούν οι εμπορικές τράπεζες και των άλλων που είναι επικίνδυνες. Μπορεί να παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο πιστεύω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από ότι τώρα με τα project bonds που αναφέρθηκαν που ελπίζω να μπορούν να προσαρμοστούν και στο μέγεθος των επενδύσεων, δηλαδή να μπορούν να προσαρμοστούν και σε μικρότερες επενδύσεις ακόμα. Ο κύριος Κόλλα από τη Σλοβακία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να ε, επενέσω την ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην ε, Σλοβακία, ιδιαίτερα σε θέματα υποδομός και δρόμων. Να συμφωνήσω επίσης σε ό,τι αφορά τους, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ευρωομόλογα, ως ένα εργαλείο για την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχεδίων. Προαπαιτείται να πληρούνται Όλη η όριση ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση, η προτινόμενη χρηματοδότηση με τη χρήση των ευρωμολόγων θα σήμαινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτούσε τις απαιτήσει αυτές όχι μόνο μέσω των ε, συνεισφορών αλλά και μέσω χρέους. Γι' αυτό λοιπόν η εισαγωγή οποιοδήποτε μηχανισμού χρηματοδότησης νέου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα περιόριζε τα ταμεία της, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις περιφέρειες που αφιερώνονται για την επίτευξη των στόχων του 2020 ή θα μείωνε τις ε, συνεισφορές των κρατών μελών. Ίσως να χρειάζονται και οι δύο μέθοδοι για μακροπρόθεσμο, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά δεν συνάδουν με τις αρχές της αλληλεγγύης και της... Ε, ο λόγος είναι ότι η εξέλιξη των διαφορών περιφερειών γίνεται πιο κεντρικός και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι η Σλοβακία υπέρ της εισαγωγής ευρωομολόγων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Άννη Ποδηματά από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να σημειώσω και εγώ από την πλευρά μου ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι απασχολεί και τη σημερινή μα συζήτηση και υπογραμμίστηκε από πολλού από του ομιλητέ, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, είναι πώ θα αντιμετωπίσουμε το, το κενό χρηματοδότηση που δημιουργεί η σημερινή κρίση ε, και πώ θα διασφαλίσουμε ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία τους μεγάλους στόχους που έχουμε μπροστά μας. Αναφέρομαι κυρίως τους στόχους που περιλαμβάνονται στη νέα μας στρατηγική για το 2020, ε, αλλά και τις άλλες μεγάλες προκλήσεις τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο ε, παγκόσμιο επίπεδο. Και ήθελα να σημειώσω, απευθυνόμενοι και προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοινός τόπος ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, από τούδε και στο εξής και λόγω της κρίσης των περικοπών στους εθνικούς προϋπολογισμούς, στον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την ε, προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Ε, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, πολύ μεγάλες δυνατότητες άντλησης νέων πόρων και το δεύτερο στοιχείο, εξίσου σημαντικό, είναι ότι ε, δεν επιβαρύνουν ε, περαιτέρω τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, σε τελευταία ανάλυση. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε ε, στην εισαγωγική σας ομιλία, στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ευρωπαϊκά ομόλογα υποδομών ε, και ήθελα να σας θέσω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Στο κείμενο διαβούλευσης που έχει δώσει στην ε, δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γίνεται λόγος για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών των, αυτών των έργων υποδομών και σημειώνεται ότι τα προσεπιλογήν έργα, τα επιλέξιμα έργα θα πρέπει ε, να είναι μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και επειδή, όπω αντιλαμβάνεστε, ε, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπω, ήθελα να ρωτήσω αν είναι προπόθεση ο διασυνοριακό χαρακτήρα αυτών των έργων, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφερθήκαμε, αναφέρθηκα και άλλοι συνάδελφοι στη στρατηγική 2020, εάν μιλάμε μόνο για έργα υποδομών ή και για πολιτικές που έχουν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την στρατηγική 2020. Ευχαριστώ πολύ. από τη Σουηδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Το θέμα τη σημερινή συζητήσεω είναι σημαντικότατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιαστεί επί τη αυξήσεω τη ανταγωνιστικότητό τη, τη αναπτύξεώ τη, εξέλιξή τη. Η αποτελμάτωση δεν αποτελεί επιλογή. Ποια μέτρα δεν αληφθούν. Καταρχάς θεωρώ σημαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Αυτό ήδη το τόνισαν πολλοί ομιλητέ. Μία ολοκλήρωση εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει τα έτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 10%. Εξυγχρονισμό και βελτιώσει απαιτούνται. Εστεζόμενοι επί τον το τομέα τη υπηρεσία και χρειάζεται και ένα πρόγραμμα ψηφιακό και γενικό σύστημα ευρεσιτεχνία και κανόνε περί απλουστεύσεω. Δεύτερον, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε όσον αφορά τις νέες στρατηγικές και την αύξηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, αλλά ό,τι και να λέμε, εάν δεν δράσουμε θα γίνει τίποτα. Πιστεύω ότι πολλά σκαλά διατυπωμένες στρατηγικές και στόχοι έχουν τεθεί. Η στρατηγική του 2020 της Ευρώπης έχει εγκριθεί και την υποστηρίζω τρόπος. Τώρα από τα λόγια πρέπει να περάσουμε στη δράση θα πρέπει να ξεχρονίσουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά να ακολουθήσουμε και κάποια περιοριστική προσέγγιση. Θα πρέπει να κατευθύνονται επενδύσει προ του νέου τομεί αναπτύξεω. Σήμερα σχεδόν το μισό του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δαπανάται επί τη κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό δεν συνάδει πλήρω με τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώση του 2020 που θέλει να αναπτύξει νέου τομεί. Θέλουμε να εξυγχρονισμό, χρειάζεται αύξηση επενδύσεων σε άλλου τομεί, όπω έρευνα, υποδομέ, παιδεία. Η λύση σε όλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι μεγαλύτερο ο υπολογισμό. Τα χρήματα του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι τα χρήματα των φορολογουμένων. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί συνετοί. Τα δημοσιονομικά θα πρέπει να είναι εξισορροπημένα. Άρα απαιτείται μεγαλύτερο σεβασμό ε, για του κανόνε και συμμόρφωση με αυτού, όπω το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Η Σουηδική Επιτροπή για τα Οικονομικά είναι κάθετα αντίθετη σε φόρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όχι, ούτε η πολιτική τη Σουηδία, ούτε ο λαό τη Σουηδία υποστηρίζει αυτό το φόρο. Κατά την άποψή μου, ο φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι κακή ιδέα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και πιο πλούσιο κόσμο και μια πιο πλούσια Ευρώπη εν κατακλείδη είναι η ώρα της δράσης ούτως ώστε η στρατηγική της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020 να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ. Τώρα τον κύριο Μποσκαριάν από τη Ρουμανία καλό να λάβει το λόγο. Δεν είναι εδώ, οπότε ο κύριος Γιάννησεν από τους φιλελεύθερους στην Ευρώπη. Η κυρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Μέιστατ για μια πολύ καλή ομιλία. Πράγματι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε. Χρειαζόμαστε τεράστιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους έχοντας εδώ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ να εκφράσω την απογοήτευση και την πίκρα που πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχηγοί κατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης, οι πρωθυπουργοί σας, συμφώνησαν επί σχεδίου δράσεως. Είναι ένα σχέδιο που αφορά την ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι τεράστιες επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν στον ενεργειακό τομέα. Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν έχουμε χρήματα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε πιει τη σαμπάνια και έχουν υποθεί αυτά, έρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών και μας λένε «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Γι' αυτό ο κύριος Μάιστα θα πρέπει να εφεύρει κάτι και θα πρέπει να βρεθούν χρήματα. Υπάρχουν προγράμματα που χρήζουν χρηματοδοτήσεις από τον προπολογισμό, όπως αναφέρατε. Υπάρχουν προγράμματα που δεν έχουν αξία τόσο υψηλή που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την αγορά. Αλλά έχω ένα παράδειγμα και για το Σλοβάκο συνάδελφο να το ακούσει. Για τα ομόλογα των έργων, τα project bonds, στη χώρα μου, τη Δανία, ε, έχουμε τεράστια κρατική επιχείρηση που επενδύει στην αιωλική ενέργεια. Και αυτή θέλει να βγει στην αγορά και συμφώνησε με κάποια συνταξιδοτικά ταμεία να δώσουν τα συνταξιδοτικά ταμεία χρήματα στο πρόγραμμα αυτό για την αιωλική ενέργεια. Είναι επίσης και ευρωπαϊκό πρόγραμμα, διότι η ενέργεια δεν θα πάει μόνο στη Δανία, θα πάει και στις βαλτικές χώρες και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Όμως, τα συνταξιωτικά ταμεία δεν μπορούν να υπομισθούν τον πλήρη κίνδυνο και χρειαζόμαστε εσά κύριε Μέιστατ να έρθετε και να χρηματοδοτήσετε το, την πολύ επικίνδυνη αυτή επιχείρηση όπως όταν έχουμε τσουνάμι το τσουνάμι που μπορεί να καταστρέψει αυτό το αιωλικό πάρκο δηλαδή κάτι που είναι απρόβλεπτο αλλά ίσως συμβεί στο μέλλον Αυτά που μας εξηγήσατε λοιπόν για τα ομόλογα των έργων, τα project bonds, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την δημιουργία αυτού του προγράμματος. Κύριε Ζιώσα από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ως εκπρόσωπος του Εγκρικού Κοινοβουλίου μπορώ και βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω ε, μπροστά σας. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Μύρο και ο κύριος Μάιστα. Ο κύριος Μάιστα δυστυχώ δεν ήταν εδώ στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης, αλλά ουσιαστικά είπαμε στην αρχή ποιο είναι ο πυρήνα τη υπόθεση, ότι δηλαδή η κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αυτό που εμείς αποκαλούμε φούσκα των ακινήτων αποτελεί μια διευθυντική κρίση του τομέα των ακινήτων. Η Ευρώπη μπορεί λοιπόν να είναι επιτυχής μόνο αν καταφέρει να αντιμετωπίσει την κρίση, την διαστατική αυτή, η οποία επικρατεί και σε εμά. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε ο κύριος Μάιστατ και θα ήθελα να πω ότι εμείς θα πρέπει να κινηθούμε και να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω. Η επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη, είπε ένας συνάδελφος. Να σας ρωτήσω λοιπόν, τι γίνεται με την προηγούμενη δεκαετία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαπιστώσουμε τη μεγάλη αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας και να φροντίσουμε να μην επαναληφθεί. Θέλουμε μια ενοποιημένη, ενσωματωμένη Ευρώπη και αυτό συνεπάγεται μεγάλα πλεονεκτήματα και στις αγορές. Πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως είπε και ο κύριος Μάιστατ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα της ταχύτητας της ταχείας λήψης αποφάσεων στην κρίση. Ευχαριστώ η κυρία Μάρτινς από την Πορτογαλία τώρα, λέει ο Πρόεδρος, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω πόσο χρήσιμο ήταν αυτά που είπε ο κύριος Μάιστα, το ότι είναι απαραίτητες οι επενδύσεις, γιατί χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχει και απασχόληση. Ωστόσο, Είπε με πάσα σαφήνεια ο κύριος Μέισταρτ ότι η ύφεση του 2009 οφείλεται στην μείωση των επενδύσεων. Άρα είναι σαφές πόσο ε, ουσιοδούς σημασίας είναι οι επενδύσεις. Είναι όμως όλες οι επενδύσεις ε, ιδιές, οι επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, οι επενδύσεις ε, σύμφωνα με την στρατηγική το 2020 οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, γιατί αυτές είναι ασφαλώς οι επενδύσεις οι οποίες ε, διασφαλίζουν μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η Πορτογαλία τον τελευταίο καιρό έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στον τομέα της ανέργειας. Έχει επενδύσει σαφώς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Πορτογαλία, σε ολική ενέργεια και υδροελεκτρική ενέργεια. Και θα θέλαμε αυτό να το υπογραμμίσουμε. Αυτό ορίζεται και από την νομοθεσία. Άρα οι επενδυτές μπορούν να προβούν σε τέτοιε επενδύσει, γιατί πρόκειται για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμε επενδύσει. Άρα είναι πάρα πολύ σωστό το γεγονό ότι ορίζονται και νομικά. το Χούμπνερ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω διευκρινίζοντα ότι αυτά που είπε ο κύριος Μάιστατ Φυσικά η χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι πάντα μια πρόκληση, αλλά και η χρηματοδότηση των στόχων του 2020 για την παραγωγικότητα, για την ανάπτυξη, για την ε, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί ακόμα πιο μεγάλη πρόκληση για μας στην Ευρώπη. Και είπατε κύριε Πρόεδρε ότι οι εθνικές περικοπές, οι περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα εξακολουθήσουν για κάποιο καιρό. Μιλήσατε για το ρόλο και των ιδιωτικών ε, τραπεζών για τους επόμενους μήνες και ίσως και χρόνια να τονίσω ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για το 2013 και μετά θα είναι περιορισμένος και ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ο ανταγωνισμός στο παγκόσμιο προσκήνιο για τα μέσα χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει να ξυπνήσουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση να τονίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέσο δημόσιου, δημόσιας χρηματοδότησης σε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο και σε εθνικό επίπεδο. Και φυσικά ο ρόλος σας ως τράπεζα και ο προσωπικός σας ρόλος είναι πιο σημαντικός παρά ποτέ. Μία έκκληση λοιπόν έχω να σας απευθύνω στο πλαίσιο αυτό. Επειδή ξέρετε και από την εμπειρία σας ότι ένας από τους λόγους που οι επενδυτές δεν προβαίνουν πρόθυμα σε νέα επενδυτικά προγράμματα είναι πολύ συχνά ότι το νομοθετικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υπερβολικά περίπλοκο. Εφιαλτικό συχνά. Για οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ελπίζω αυτά τα project bonds, τα έργα υποδομών να, για τα έργα υποδομών να είναι πιο εύκολα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εργάζεται και ξέρω ότι και εσείς συμμετέχετε στην εργασία αυτή για μια νέα νομοθεσία. Να σας ζητήσω λοιπόν να φροντίσετε να είναι πραγματικά καλό το ρυθμιστικό πλαίσιο, να βελτιώσουμε πραγματικά το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο σε πολλούς τομείς θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία καταρτίζεται. Θα, θα χρειαστούμε λοιπόν συγκεκριμένους όρους για τον έλεγχο, για την... Ε, τον ορισμό των σχετικών όρων. Εκ των προτέρων θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά και θα πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα... Ναι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, θα πρέπει να σας διακόψω. Ναι, με ολοκλήρωσα λέει η ομιλήτρια. Ο κύριος Στούνφολ από την Αυστρία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτά που συζητούμε εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις και η επιτυχία ή η αποτυχία θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό και νομίζω ότι η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 αποτελούν εξαιρετική βάση αλλά δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της στρατηγικής Λισαβόνας όπου ενθουσιαστήκαμε με τη ρητορική και μετά δεν μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε. Έχουμε μία μοναδική δυνατότητα να επιτύχουμε εάν οι βασικοί στόχοι της ε, στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 ε, ενταχθούν και στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και αυτό κάνουμε στην ε, Αυστρία για την οικονομική μας πολιτική. Όσον αφορά για το μέλλον, νομίζω ότι η προτεραιότητα των επενδύσεων πρέπει να είναι οι στόχοι μας, η οικονομία, η παιδεία, η υγεία, οι κοινωνικές δομές, αλλά ε, ποιος ε, μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης των εξωτερικών παραγόντων της Κίνας, της Ινδίας, μόνο οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρέπει να βρεθούμε σε μία θέση παγιδευμένη μεταξύ των Ανατολών με την Κίνα και την Ινδία και δυσμών με τις Ηνωμένε Πολιτείες και να μπορέσουμε ε, να ε, θεωρήσουμε ότι η στρατηγική μας για το 2020 θα μπορέσει να μας βοηθήσει βάσει συζητήσεων που δεν θα γίνονται μόνο μια φορά το χρόνο αλλά πιο συχνά. Ο κύριος Βαντάλ τώρα έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ε, μιλώ εξ ονόματος του κόμματος ε, για την ελευθερία. Η, Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη εξέρχεται σιγά σιγά από την κρίση και ανησυχούμε ιδιαίτερα για το μέλλον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση, αλλά το θέμα είναι ασφαλώς πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία και την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα να ε, φροντίσουμε και τα δημοσιοοικονομικά μας και να θέσουμε και πιο αυστηρούς κανόνες για τις τράπεζες. Το κόμμα μας ανησυχεί για θέματα ε, κυριαρχίας των κρατών μελών. Για εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πολιτική ένωση και δεν θέλουμε ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό υπερκράτος και φαίνεται ότι όλα καθίστανται πιο ρευστά και ότι αυτή η κρίση όλο και οδηγεί σε μια πολιτική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί τα κρατημέλη και όχι αντίστροφα και το ΠΒΒ, το κόμμα μας, θα είναι πάντα αντίθετο σε τέτοια ε, παραχώρηση των εθνικών αρμοδιοτήτων και κατά οποιασδήποτε μορφής ε, φορολογικής ε, ευρωπαϊκής φορολογίας. Είτε μιλάμε για ευρωομόλογα, είτε για ομόλογα αργά υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει φορολογική αρχή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνέρχονται και να ακολουθούν το ισχυρότερο κράτος μέλος και όχι αντίστροφα. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο αδυναμός κρίκος και θα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Οι χώρες έχουν την ε, ευθύνη τους και θα πρέπει να καταστούν ε, ανταγωνιστικές. Δεν το ακούω αυτό σήμερα. Φαίνεται λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται υπεύθυνη για να καταστήσει τα κράτη μέλη ανταγωνιστικά. Αντολίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η στρατηγική του 2020 αναφέρθηκε και όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε επενδύσεις σε ένα κλίμα γενικής α, ε, λιτότητας έχει, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες διότι για την ώρα οι προσπάθειες γίνονται για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα ελλείμματα, να βελτιώσουμε την ποιότητα των επενδύσεων κλπ. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα αποθέματα. Αυτές οι προσπάθειες που καταβέλλονται τώρα. Η στρατηγική για το 2020 απαιτεί να κάνουμε κάτι για το έλλειμμα στις επενδύσεις. Χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές, χρειάζονται επενδύσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, στα ενεργειακά δίκτυα, ε, όπως είπε και ο πρόεδρος Μαϊστάντ. Είπε ένα 1,5 με 2 ε, δις. Ε, σχεδόν δύο φορές οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δύο-τρεις μάλλον χρειάζεται να επενδύσουμε και επί της παιδείας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα βρεθούμε στη δυσχερή θέση. Στη Φιλανδία υπολογίστηκε ότι πάνω από ένα με δύο εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται κατά άτομο για τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτοί που δεν έχουν τη σωστή παιδεία τελικά καταδικάζονται στην ανεργία. Θα πρέπει να επενδύσουμε και στην έρευνα και την νέα τεχνολογία και θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να, φε... να φέρνουμε και το ταλέντο, να προσελκύουμε και το ταλέντο από το εξωτερικό. Οι μετανάστες εξειδικευμένοι δεν είναι στους αριθμούς ε, που είναι στη ΣΥΠΑ και είναι το ένα πέμπτο από αυτούς τους εξειδικευμένους που πάνε στην Αυστραλία και το ένα τέταρτο από αυτούς που πάνε στον Καναδά. Χρειάζεται τριπλή προσέγγιση. Αντίθετα από τους άλλους ομίλητες, εγώ νομίζω ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα. Θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος του συστήματος και το ποσοστό της εθνικής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί φυσαλίδες οικονομικές, αλλά τα χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία. Άρα χρειάζεται πολύ βαθιά οικονομική μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση του προπολογισμού. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν αρκούν, άρα θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να προσελκύσουμε και άλλες επενδύσεις. Αναφέρθηκε ο φόρος των χρηματοστοτικών ε, συναλλαγών και το πρασίνισμα της οικονομίας. Αλλά χρειαζόμαστε ανακατανομή του φορολογικού βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι που θύμισε ο κ. Μέιστατ, ότι χρειάζονται επενδύσει για την καινοτομία, για τη διάδοση τη καινοτομία, για τον μερισμό των κινδύνων. Χρειαζόμαστε και τα project bonds. Σα τελείωσε ο χρόνο, λέει ο πρόεδρο Δικόπτη. Χρειαζόμαστε συντονισμένε ευρωπαϊκέ επενδύσει. Και αυτό. Εάν δεν συντομεύεται, τελειώσουμε Ε, και έχουμε ακόμα μισή ώρα, έχουμε μακροσκελή κατάλογο. Να δώσω και το λόγο και στον κύριο Μάιστατ και στου ε, εισηγητέ να συνοψίσουν. Αντροκάητη από την Λιθουανία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Αντρουκάιτης. είναι πολύ καλό, θα ήταν καλό να έχουμε ένα ξεκάθαρο κανόνα. Να έχουμε μια θεώρηση των πραγμάτων ε, σφαιρική, να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται στον κόσμο και να κινούμεθα και στο τοπικό επίπεδο. Έχουμε 27 εθνικά κοινοβούλια που παρίστονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται συντονισμό των δράσεών μα για να πετύχουμε του στόχου μα για το 2020. Αυτό που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει σχέσεις μεταξύ του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των μακροοικονομικών μέτρων αυτού με τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Θα πρέπει να συντονίσουμε αυτή τη διασύνδεση. Η Λιθουανία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Το Κοινοβούλιο μας υιοθέτησε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά το εξάμεινο της Προεδρίας αλλά πρέπει να προσέξουμε και αυτή την πτυχή και η περιφερειακή συνεργασία το χώρο της Βαλτικής είναι ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Διάφορα προγράμματα στην περιοχή μπορούν να συνδέσουν τα κράτη της Βαλτικής και όλη τη Βαλτική θάλασσα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα ευρωμόλογα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ για την εκτέλεση των μέτρων και των έργων. Τα ευρωμόλογα λοιπόν θα επιτρέψουν να υλοποιήσουμε καλύτερα τα έργα προγραμματίζουμε και στην περιοχή μας. Η, στα, η στατική για τη Βαλτική σήμερα πιστεύω ότι θεωρείται εξαιρετική. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία Ντελόρ Μπούζεκ να συναυθεί σήμερα αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη, συντονισμένη δράση. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γένσεν. Θα, Μπένσεν, θα συνεχίσω στα δανέζικα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Φιλίπ Μάιστατ για τα όσα μας είπε. Ήταν έξοχη η εισαγωγή που έκανε. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε όσον αφορά την μακροπρόθεσμη δανειοδότηση, χρηματοδότηση της τράπεζας. Ε, στο μέλλον θα είναι περιορισμένη η χρηματοδότηση από και υπάρχουν και δημοσιονομικέ δυσκολίε σε διάφορα κράτη-μέλη και θα συνεχιστούν αυτέ και τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι το σύστημα των εγγύσεων που έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο για να εξευρεθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για τους στόχους του 2020. Αυτοί οι στόχοι λοιπόν μας βρίσκουν συμφώνους. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε τάξη στα του οίκου μας πρώτα απ' όλα. Περνάμε μια οικονομική κρίση, μια χρηματοπιστωτική κρίση και θα πρέπει τώρα να προσελκύσουμε τις επενδυτές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουν πίστη στις οικονομίες των διαφόρων χωρών οι επενδυτές. Και το θέμα είναι, έχουν εμπιστοσύνη. Όχι. Υπάρχουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχουν δαπανίσει περισσότερα από αυτά που κέρδισαν. Ζήσαμε πέρα από τα όρια μας και τις δυνατότητές μας και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε έκδοση ομολόγων ε, κρατικών πολλών ε, δημιουργήθηκε κρατικό χρέο μεγάλο και έχουμε το πρόβλημα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ασία. Ας μην αναμειγνύουμε τα πάντα βέβαια. Εμείς είμαστε σε κάποια παγίδα πολυτελή αν θέλετε. Ε, ε, έχουμε ψηλούς μισθούς, μεγάλες διακοπές. Ζούμε σε ένα κλουβί χρυσό και προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως είναι της Ασίας. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν. Εγώ συμφωνώ με τα ευρωομόλογα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλε μορφές για την αγορά εργασίας. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πρέπει να βελτιώσουμε την αγορά εργασίας μας. Δεν συμφωνείτε επίσης, κύριε Μέιστατ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις με τα συστήματα που υπάρχουν και γνωρίζει. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θα είναι δύσκολο να απαντήσω σε ένα λεπτό. Καταρχήν όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μέιστατ εάν υπάρχει συσσόρευση ή απλώς λογικές υποδομές διότι μιλάμε για το φυσικό αέριο έχουμε τρία δίκτυα είναι λογικό διασύνδεση ηλεκτρικού πρέπει να υπάρχει διασύνδεση ή να υπάρχει αποκεντρωμένη διανομή ηλεκτρικού στις διάφορες περιοχές και ε, για την πράσινη ανάπτυξη. Μετά από αύριο θα υπάρχει η ίδια. Δεν μιλήσατε για την έρευνα, αλλά νομίζω ότι και αυτή είναι σημαντική επένδυση. Και τέλος, επειδή έχω ελάχιστο χρόνο, δύο-τρία πράγματα ακόμη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο ε, πρεσβεύεται είναι ε, πολύ εντυπωσιακό ότι μόνο το δημόσιο μπορεί να αναλάβει ε, τους κινδύνους εδώ αναφέρομαι ε, στις τράπεζες και για τη Βασιλεία 3 νομίζω ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις τράπεζες ε, των οποίων, ε, οποίων αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση από ότι εις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις πατάλες και ιδίω του δημοσίου τομέα θα ήθελα να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε και τις ιδιωτικές ε, σπατάλες οποίες δεν αναφέρεται. Περβόνς, αντιλαμβάνουμε θέλετε να κάνετε μία ερώτηση στον κύριο Μάιστερ. Θα το συνδυάσετε με την περίληψή σας. Ίσως όχι. Η ερώτηση μου είναι ταχύτατη. Δηλαδή, όσον αφορά την θεώρηση των επενδύσεων και την δυσκολία να εξεύρουμε τις ενδεδειγμένες επενδύσεις ε, είναι ένα βασικό θέμα στην Επιτροπή Κρίσης που εξετάζουμε. Αλλά πώς αυτοί οι νέοι τρόποι καινοτόμων χρηματοδοτήσεων μπορεί να κινητοποιήσουν την αποταμίευση των Ευρωπαίων και ε, όχι ε, μόνο των ε, κυριάρχων ε, κεφαλαίων των τρίτων χωρών και πώς αυτά τα μεγάλα προγράμματα υποδομής λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσει συνοχής και συγκλήσεως, το οποίο ήταν ένας από τους λόγους κρίσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κύριε Μάιστατ, τώρα έχετε το λόγο για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα τα σχόλια, σε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα υπάρξουν πάλι οι συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες οι οποίοι θα τοποθετηθούν ένα-δύο λεπτά. Ξεχάσαμε όμως κάτι. Πριν δώσουμε το λόγο σε εσά, πρέπει να μιλήσει ο κύριος Τσιρόνης από την Ελλάδα, ο οποίος είχε εγγραφεί και τον ξέχασα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να μετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις με συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των Εθνικών Συμβουλίων των Κρατών Μελών. Οι στόχοι των κρατών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, να ικανοποιήσουν από τη μία πλευρά την ανάγκη για χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μείωση των ελλημάτων και το χρέους τους και από την άλλη πλευρά την ανάγκη για ανάπτυξη και συνοχή είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων αντικρουόμενοι και τελικά οι οικονομίες τους υποφέρουν από ύφεση, ανεργία, φτώχεια, κοινωνικό εξοπλισμό και τελικά αύξηση των χρεών του. Ε, απαιτούνται επιπλέον πόροι για την χρηματοδότηση τη ανάπτυξη και τη συνοχή και την αντιμετώπιση τη κρίση αυτών των χωρών. Η Ελλάδα υποστηρίζει αυτή την ανάγκη αύξηση των πόρων τη συνοχή και τη ανάπτυξη και στην κατεύθυνση αυτή ήταν και η αποφάση του πρόσφατου άτυπου Συμβουλίου Κορυφή για, τον μόνιμο μηχανι... Ε, για το μόνιμο μηχανισμό σταθερότητα που αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Ε, τα νέα χρηματοδοτικά επίση εργαλεία που ανέφερε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι απλά, κατανοητά και αποτελεσματικά, που θα βοηθούν του στόχου τη ανάπτυξη και τη συνοχή, κατευθύνοντα του πόρου στην πραγματική οικονομία και όχι στην κάλυψη των ρίσκων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Ελλάδα πιστεύει ότι θα πρέπει να εισαχθεί η περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά την επιλογή των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, Θεωρούμε επίση ότι ο πολιτισμό και ο τουρισμό που δεν αποτελούν επιλεγμένη προτεραιότητα πρέπει να βρουν τη θέση του στη νέα προγραμματική περίοδο, όπω και ο πρωτογενή τομέα που η συνέχιση τη ενίσχυσή του αποτελεί προτεραιότητα. Τέλος, η εδαφική διάσταση αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής συνοχή για την Ελλάδα και προτείνουμε να εξεταστεί ενίσχυση και αναβάθμιση του στόχου 3 της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, με την ενσωμάτωση των περιοχών με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπω είναι οι νησιωτικές περιοχές, καθώς και οι ουρινέ και απομονωμένε περιοχέ. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχετε το λόγο, κύριε Μάιστατ. ο πρόεδρος μου δίνει ελάχιστο χρόνο, οπότε παρακαλώ εκ των προτέρων να, ε, να με συγχωρήσετε, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα ενδιαφέροντα σχόλια που άκουσα. Θα επικεντρωθώ σε τρία θέματα που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Καταρχήν ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι βασικές για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απασχολούν κάτω των 250 ατόμων και εκεί εστιάζεται ουσιαστικά η απασχόληση. Άρα και πολύ σωστά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτή τη διάσταση Κατόπιν όμως αιτήσεως των μετόχων μας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση προς τις τράπεζες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα βρείτε τα στοιχεία στο σημείωμα που έχει κατανεμηθεί και τώρα μπορούμε καλύτερα να παρακολουθήσουμε την ουσιαστική και πραγματική χρήση αυτών των κεφαλαίων για να δούμε αν οι τράπεζες όντως βελτιώνουν την πρόσβαση στην, ε, στις πιστώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή όχι. Πολύ σωστά είπε η κυρία Πιτικέινεν προηγουμένως ότι δεν υπάρχει μόνο το θέμα των πιστώσεων αλλά και τα κεφάλαια κινδύνου όπου πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε ένα ε, τμήμα το οποίο ασχολείται με τέτοια κεφάλαια που συμμετέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυξήσαμε τις δυνατότητες του υποκαταστήματός μας σε αυτό το θέμα και υπάρχει και το πρόγραμμα SIP της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συμβάλλει επίσης εις ε, τις περισσότερες δυνατότητες χρηματοδοτήσεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, είμαι πολύ γενι... Ε, μιλώ σε πολλές γενικές γραμμές, συγχωρήστε με, αλλά μπορούμε να εμβαθύνουμε μετά τα θέματα αυτά. Μετά, το θέμα του προγράμματος των ομολόγων, διότι υπάρχουν ακόμη παρανοήσεις. Ο πρόεδρος Ντολόρας με, ας με συγχωρεί, αλλά όταν μιλώ στους δημοσιογράφους για τα ομόλογα αυτά, ε, διαφοροποιώ μεταξύ τα Delors bonds, τα Juncker bonds και τα Barroso bonds, δηλαδή τα ομόλογα Juncker, Barroso ή Delors. Εγώ είμαι υπέρ και των τριών, αλλά είναι τελείως διαφορετικές δυνατότητες. Τα ομόλογα Delors είναι ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε επίσης να δανειστεί για να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές ε, και επενδυτικές δαπάνες ε, το οποίο ήταν μια ιδέα του Προέδρου Ντελόρ ε, για να χρηματοδοτήσουμε τα δίκτυα ενεργείας και μεταφορών διότι και πρέπει να το παραδεχθούμε έτσι αυξάνουμε το χρέος Ευρωπαϊκής Ενώσεως πράγμα το οποίο πολύ ορθόδοξο δημοσιονομικά εφόσον απλώς ε, δανειζόμασταν για να χρηματοδοτήσουμε ε, την, ε, την ανάπτυξη που αύξανε την συλλογική περιουσία. Αυτό ήταν το πρώτο είδος. Το δεύτερο, τα ομόλογα Juncker, είναι ε, μία αμοιβαία ευθυνή για ένα μέρος των χρεών των κρατών μελών. Μπορεί να γίνει με, ε, κατά κάποιον τρόπο αμοιβαία κεφάλαια ή αμοιβαίες υποχρεώσεις των κρατών μελών με κοινά χαρακτηριστικά ώστε ένα μέρος του χρέους και είναι, υπάρχουν τέτοιες προτάσεις να μπορούμε λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε με αμοιβαία κεφάλαια ένα μέρος με αυτά τα ομόλογα από τις επενδύσεις μας και υπάρχουν και τα ομόλογα Μπαρόζο που ο εκδότης δεν θα είναι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τα κράτη-μέλη αλλά μία εταιρεία που θα αναλαμβάνει το πρόγραμμα είτε ιδιωτική είτε μεικτή ιδιωτική και δημόσια και αυτή θα καταρτίζει τα προγράμματα και θα εκδίδει τα ομόλογα αλλά θα πρέπει να υπάρχει το επίπεδο ποιότητος που θα επιτρέπει σε θεσμικούς επενδυτές να τα αγοράσουν. Είπα λοιπόν στον κύριο Βέμπερ ότι ε, δεν πρέπει όλος ο κίνδυνος να αναλυφθεί από το δημόσιο τομέα αλλά απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους επενδυτές οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα γιατί αυτό που χρειαζόμαστε για τα προγράμματα αυτά είναι μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και πρέπει να στραφούμε προς τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν δεσμεύσεις και μπορούν να επενδύσουν μόνο σε χρεόγραφα τα οποία έχουν ε, εξαιρετική βαθμολόγηση α και ενδεχομένως 2α και αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα του προγράμματος. Πάντοτε υπάρχουν κίνδυνοι για τα προγράμματα υποδομής. Άρα ε, θα πρέπει να επιτύχει αυτό το χρεόγραφο μία εξαιρετικά καλή βαθμολόγηση. Γι' αυτό και εκεί μπορεί να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το καλύτερο παράδειγμα ήταν αυτό που ανάφερε η κυρία Γέντσεν για, τις, ε, για αιωλικά πάρκα, το οποίο ακολουθεί ακριβώς τη στρατηγική 2020, ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, αλλά με τέτοιο κίνδυνο που όπως το είπε πολύ σωστά, οι τράπεζες οι εμπορικές διστάζουν να χρηματοδοτήσουν και άρα θα, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια ομόλογα. Και το τρίτο θέμα, στο, το οποίο θα θίξω εντάχει αλλά είναι ουσιαστικότατο, είναι η σύγκριση που έγινε από πολλούς ε, από εσά με τη στρατηγική της Λισαβόνας που είπαμε ότι απέτυχε. Γιατί, διότι στρατηγική ε, και γιατί λοιπόν θα επιτύχει καλύτερα η στρατηγική του 2020. Δεν είναι τόσο η μορφή της στρατηγικής που δεν διαφέρει τόσο, η διάγνωση της Λισαβόνας ήταν σωστή. Ο τρόπος ε, που θα την εφαρμόσουμε είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομικής δεν θα επεκταθώ, αλλά στις συζητήσει που γίνονται τώρα και αύριο το πρωί το ΕΚΟΦΗΝ θα συζητήσει τη θέση της Ευρώπης για την οικονομική διακυβέρνηση και υπάρχουν δύο κινήσεις απαραίτητε. Αφενός πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της διακυβέρνηση καταρτίζοντας ένα μηχανισμό ε, κυρώσεων που θα είναι πιο αξιόπιστος και ελπίζω ότι θα υπάρχει και ένας μηχανισμός κινήτρων που θα υποκινήσει τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν ε, στις μακροπρόθεσμες ε, ε, προβολές αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε επίσης γιατί μέχρι στιγμής συγκεντρωνόμαστε ιδίως στα δημοσιονομικά θέματα και ο πρώην υπουργό Οικονομικών αναγνωρίζω τη σημασία του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές της οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει να συντονίσουμε. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε αν είχαμε χρόνο στο θέμα της έρευνας γιατί οι επενδύσεις στην έρευνα θα είναι πιο αποτελεσματικές αν είναι πιο συντονισμένες και για να τις συντονίσουμε πρέπει να δεχθούμε ότι πολυμερώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιοριζόμαστε μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε μακροοικονομικές θεωρήσεις. Με συγχωρείτε που ξεπέρασα την ώρα μου αλλά καταλαβαίνετε ότι πιστεύω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα θα επιτύχουμε τις στρατηγική του 2020. Τώρα καλώ τους πέντε συντονιστές και θα παρακαλούσα ο καθένας να μιλήσει πέντε, ένα λεπτό για να έχει υπερβόνσο ακόμη πέντε λεπτά στο τέλος. Ε, ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Ιστορική υπενθύμηση. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα υπάρχουν από το 1953. Οπότε υπήρξε ε, ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής Συνθήκης που δυστυχώς ποτέ δεν υιοθετήθηκε όπου έλεγε το ότι ε, τα ευρωπαϊκά ομόλογα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν είναι τόσο επαναστατικό. Ένα νέο στοιχείο που μας ε, παρουσίασε ο πρόεδρος Μάιστατ τα 15-20 δισεκατομμύρια για την έρευνα ε, μέχρι ε, το 2020 αντι ε, προσωπεύουν 10 έως 20 εθνικούς προϋπολογισμούς, άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ευρωπαϊκά εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο επίπεδο των αναγκών μας για να μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε και δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει μία πλήρη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών συστημάτων. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη επιχειρήσεων, έχουμε ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ευρώπη οι οποίες φτάνουν σε ένα κρίσιμο μέγεθος για να μπορέσουν να αντιταχθούν και να ανταγωνιστούν ξένες και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο κινδύνου. Και αν δεν μπορεί να έρθει ευλόγως από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να προέρθει είτε από δημόσιες πηγές ή από, το δημόσιο, από ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ανησυχώ από το διαχωρισμό που κάνουμε στη συζήτησή μας. Ποιο διαχωρισμό μεταξύ των ειδικών τομέων που, για τον οποίο δεν έχω παρατήρηση όσον αφορά το πικιος Μάιστατ που αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 από τους όρους του γενικού πλαισίου από την άλλη. Ακούσαμε και σήμερα ότι πολλοί είναι πεπισμένοι και εγώ μένω από αυτού, ότι χωρίς μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί το ευρώ αλλά χωρίς το ευρώ ε, δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική για το 2020 που θα εφαρμοστεί σωστά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό συνεπώ να φροντίσουμε το ώστε κάθε φορέας, θεσμική εκπρόσωπη, πολιτική, κοινωνική φορείς να έχουν μια, ε, κάποια κυριαρχία ε, αλλιώς θα πετύχουμε το στόχο μας. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Η υλοποίηση των μέσων, όπως αυτός που, εγγυα, εγγυάται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να, να, να είναι εκτός τελικά των θεσμών της, της Ευρώπης. Έχουμε ε, διτή προσέγγιση, έχουμε χρηματοδότηση νόμως από τη μία πλευρά ε, και από την άλλη πλευρά θέλουμε τις παρεμβάσεις για την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ, Όλη Σμίτ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη η συζήτηση. Δεν μιλάμε για την απαρχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, μην το φοβάστε αυτό. Όχι, συζητάμε, μιλάμε για την αρχή μιας συζήτησης όπου όλοι από τις χώρες μας και για τους πολίτες που, που εκπροσωπούμε εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά το γεγονός ότι πολλοί ότι υπάρχει σεβασμός για την άποψη ότι κάποιοι θεωρούν ότι η Ευρώπη που έχουμε στα χέρια μας είναι πολύ λίγη. Όπως και να έχει, εξαρτώμαστε από ένας από τον άλλον με τρόπο που δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε πριν από 5-10 χρόνια. Δύο σχόλια. Ο Λόρδος Λίντον Χάρισον. Ήταν πολύ καλό το ότι μας είπατε ότι σκέφτεστε στα εμπορίου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν ένα Ηνωμένο Βασίλειο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την προστασία της ενιαίας αγοράς. Κύριε Φαντέικ από την Ολλανδία, να σας πω ότι ασφαλώς μπορεί να είσαστε επικριτικοί, αλλά δεν υποτίθεται ότι μπορείτε να κατηγορείτε την Ευρώπη για ό,τι συμβαίνει. Να είσαστε επικριτικοί, αλλά να μην κατηγορούμε τις Βρυξέλλες για τα πάντα. Γιατί αυτό το θέμα, αυτό, αυτές οι κατηγορίες ε, θέτουν και αμφισβητούν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο Ρόμπερτ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μάιστατ για την εξαιρετική του εισήγηση για τον τρόπο χρηματοδότησης ε, των υποδομών του μέλλοντος. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε νέα μέσα και ίσως ε, τα ομόλογα μπαρόσο να είναι μια καλή λύση για σε άλλες περιπτώσεις δεν, μπορούμε να, δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα TNT των διευρωπαϊκών δικτύων με δεκάδε ε, εκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν ασφαλώ, αλλά αναρωτιέμαι και ανησυχώ, επειδή στην περίπτωση αυτή θα ήταν ένα project με βάση τις ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτές, ε, αυτά τα σχέδια τα πιο επικερδή θα είναι προτεραιότητας σε ό,τι αφορά τα ομόλογα αυτά. Και τι γίνεται με το ερώτημα της ε, Περβάνς με την ιδέα της ε, συνοχής. Γιατί τα ομόλογα για έργα υποδομών θα ήταν πιο ενδιαφέροντα, για παράδειγμα, στους επενδυτές, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, Βαλτική, για τη μεγαλύτερη παροχή αερίου και για τα επικερδή φυσικά σχέδια. Ευχαριστώ πολύ ο Νικόλαος. Θα ήθελα σύντομα να πω ότι ενδιαφέρουσα η εισήγηση που μας έκανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων αλλά στη συζήτηση που ξεκίνησε ότι όλα αυτά γίνονται προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της, του 2020 ετέθη το ερώτημα γιατί απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας. Βέβαια στο τέλος από τον πρόεδρο άκουσα την εκδοχή του με την οποία δεν συμφωνώ αλλά είναι ένα κρίσιμο θέμα. Γιατί απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας ενώ ήταν καλή στη ρητορική. Και νομίζω ότι και η στρατηγική για το 2020 θα αποτύχει διότι στηρίζεται στο αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό σύμφωνο σταθερότητας που μάλιστα κατά την απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος ενδεχομένως και αυτό συμφωνεί ότι πρέπει να είναι και πιο αυστηρό να έχει και κυρώσει τα κίνητρα δεν τα βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, εξ αυτού του βασικού λόγου, κατά την εκτίμησή μου, θα αποτύχει η στρατηγική, διότι αυτό το σύμφωνο δεν είναι ότι χαλάρωσε και δεν το εφαρμόζανε, δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν ούτε οι μεγάλες χώρες και πριν από την κρίση. Δεύτερη παρατήρηση είναι συμφωνούμε με, να αναζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέα χρηματοοικονομικά μέσα, ευρωμόλογα ειδικά ο σκοπού, φόρος ε, επί των ε, τραπεζικών συναλλαγών, αλλά θα ήταν καλύτερο να επιδιώξουμε κάτι πιο σταθερό που δίνει και σταθερότητα στο ευρώ, δηλαδή αυξημένο κοινοτικό προπολογισμό και διαφορετικό ρόλο τη Κεντρική Τράπεζα. Και τέλο, δεν ξέρω αν έχει το περιθώριο να μου απαντήσει ο κύριο Πρόεδρο επί του πιο συγκεκριμένου θέματο, αν, αν, αν η Τράπεζα ανάμεσα στα άλλα έχει σκοπό να κλείσει ανισορροπίε, ανισοτιμίες στο επίπεδο της ή είναι στην επιλεξιμότητά τη Τράπεζα οι πιο αδύνατε χώρε. Δεύτερο, είναι, γιατί κάποια στιγμή δεν το κατάλαβα καλά. Λέει, επενδύσεις που δεν έχουν κέρδος είναι σπατάλη. Η επένδυση στην παιδεία και στην έρευνα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις δεν θεωρείται σπατάλη. Ναι, και τελειώνω. Μεσολαβεί η Τράπεζα Επενδύσεων μεταξύ του κοινοτικού ή και του εθνικού ε, προϋπολογισμού και του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών. Έχει εμπειρία ε, ότι σε μια ε, τέτοια περίπτωση ανεβαίνει το κόστος του έργου κατασκευής όταν εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας. Επομένως έχουμε σπατάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε ότι ο κύριος Μασιστάτη δεν μπόρεσε να απαντήσει στις δύο ερωτήσεις για την κινητοποίηση της αποταμίευσης των οικοκυριών μακροπρόθεσμα αντί να έχουμε μείγματα ή για το θέμα της συνοχής που συμφωνώ εν μέρη με αυτά που είπε ο συνάδελφος Τσίλε αλλά θα το δούμε ίσως μετά εγώ μετρώ την ευθύνη όλων σε αυτό το σημείο της συζήτησης διότι όλοι θυμούνται σαν ε, έναν εφιάλτη την αποτυχία της στρατηγικής Λισαβόνας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεκινήσουμε από την αρχή. Άρα το να δημιουργήσουμε και να επινοήσουμε νέους τρόπους χρηματοδοτήσεως αυτής της στρατηγικής μας ικανοποιεί, αλλά δεν ε, αρκεί όπως είπε από την αρχή ο Πρόεδρος. Άρα πρέπει να καταλήξουμε στα συμπεράσματα ε, για τις τις συζητήσεις που έχουμε εκ του παραλίλου και εγώ δεν θέλω να επέμβω αλλά με γνωρίζει ο πρόεδρος, τον προκαλώ κάπως στη συζήτηση και δεν μπορούμε να λέμε ότι απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας ενώ έθετε το ερώτημα της παιδείας, της γνώσης σαν α και ω της επιτυχίας της και παρακολουθούσε όχι σύμφωνα με τους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία δεν κάνει ανακεφαλαίωση των συνδρομών των προϋπολογισμών που εσείς ψηφίζετε για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εχθές της Λισαβόνας σήμερα της στρατηγικής για το 2020 και μόνο σα και οι αριθμοί του σας λέγουν ότι τα 10 χρόνια πρώτης κρίσεως το ίμιση των κρατών μελών μείωσαν τον προπολογισμό τους ε, στο θέμα της παιδείας και κανείς δεν μιλά για κυρώσεις από αυτού προς τις χώρες που μείωσαν αυτούς τους προπολογισμού, οι οποίες ευθύνονται και για το δικό τους μέλλον και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο διεθνή ανταγωνισμό. Οπότε σκεφτείτε το εξή. Εάν δούμε την νομοθεσία που καταρτήσαμε για τις τράπεζες και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, λόγω των απαιτήσεων για ίδιους πόρους τότε ε, ε, έχουμε εισάγει μεταβλητές ως προς τη φύση των ιδίων πόρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου επίπεδου για τους εμπειρογνώμονες και τις μόνες δαπάνες που αποτιμούμε διαφορετικά ή κοιτάζουμε διαφορετικά ποιοτικά είναι η συντάξεις με κεφαλαιοποίηση και νομίζω ότι αυτό είναι μια ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να γίνει για τον τρόπο με τον οποίο να μορφώνουμε το σύμφωνο σταθερότητος αφενός και δεύτερον επί των ε, επιπτώσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη νέα περίοδο προγραμματισμού που μας αφορά και σας και εμάς και ο πρόεδρος Μέιστατ ε, μας έδωσε ένα μήνυμα διότι ο μοχλός τον οποίο αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σε ένα θέμα στην πολιτική συνοχής γιατί ξέρουμε ότι ο ο εντολέας ο πιο αποτελεσματικός για τις δημόσιες δαπάνες είναι οι περιφέρειες και οι περιοχές όπου το φαινόμενο του μιουχλού για να χρηματοδοτήσουμε τη συνοχή και για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα αυτό ε, απαιτεί μία προπτική των δημοσιονομικών προπτικών διαφορετική από αυτήν την οποία να ακολουθούμε τώρα. Και θα πω μία φράση ακόμη μόνο κύριε Πρόεδρε. Σε κάθε κράτος μέλος οι κυβερνήσεις θα έρθουν να σας επισκεφθούν και να σας πούν ότι δεδομένων των εσωτερικών μου δημοσιονομικών δεσμεύσεων δεν μπορώ να αξίσω τη συμμετοχή